Συνάδελφοι, καλημέρα σας. Ας ξεκινήσουμε τη συνεδρίασή μας με την έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Εγκρίνεται. Ευχαριστώ. Περνάμε στο σημείο 2. Ανακοινώσεις του Προέδρου. Έχω μερικές ανακοινώσεις, αλλά θα είμαι πάρα πολύ γρήγορος. Ενημέρωση για τους εξέλιξη τριμερείς διαλόγους. Επιτέλους αρχίζουμε να προχωρούμε. Άρχισαν πάλι οι εργασίες τριμερούς διαλόγου να σας ενημερώσω για το πώς έχουν τα πράγματα. Στον τριμερή διάλογο για τις ευρωπαϊκές στατιστικές, ο οποίος είχε διακοπεί τον Φεβρουάριο, γιατί η εντολή που είχε ανατεθεί στην ελληνική προεδρία τότε δεν επέτρεπε να γίνει πρόοδος, τώρα συνεχίζεται. Χάρη στις επαφές που έκανε η Ιταλική Προεδρία. Οι διαπραγματεύσεις θα ξαναρχίσουν και ο πρώτος γύρος προβλέπεται στις 18 Νοεμβρίου, από τις 9 στις 12. Νέος εισηγητής είναι ο κύριος Ιγκ Μπαγιέ, και οι πολιτικές ομάδες έχουν ορίσει τους σκιώδεις εισηγητές τους για το ΕΛΚ. Η κυρία Γκαλπέλτ, για τους συντηρητικούς και μεταρρυθμιστές, ο κύριος Ότσοκ, για τους φιλελεύθερους η κυρία Ιντβελτ, για την Γκουε η κυρία Λόπες και για τους πρασίνους ο κύριος Λάμπερτ. Άλλος τριμερής διάλογος, ο κανονισμός ΕΛΤΙ, κανονισμός δηλαδή για, τις, για τα Ταμεία Μακροπρόθεσμων Επενδύσεων, Ήδη ξεκινήσαμε, ξανάρχισαν οι διαπραγματεύσει και είχαμε δύο τριμερείς διαλόγους τον Οκτώβριο και στις 5 Νοεμβρίου. Πρέπει να πω ότι υπάρχουν ε, κάποια θετικά βήματα. Οπότε προβλέπεται ο επόμενος γύρος για τις 26 Νοεμβρίου στο Στρασβούργο και μπορεί να χρειαστεί και άλλη μια συνεδρίαση τον Δεκέμβριο. Όμως έχουμε πολλές προσδοκίες, ας το πω έτσι, για τον επόμενο γύρο στο Στρασβούργο και έχω την ελπίδα ότι θα μπορέσουμε, την πεποίθηση μάλλον, θα μπορέσουμε μέχρι το τέλος του χρόνου να κλείσουμε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Αν όλα πάνε καλά, γιατί κάποια πολιτικά ζητήματα βεβαίω παραμένουν κρέμα και εφόσον επιληθούν ε, ε, γέρο. Η διπραγματευτική ομάδα είναι η εξή για το ΕΛΚΟ, κύριο Λαμασούρ, για, για τους συντηρητικούς και για τους ε, σοσιαλιστές, ο κύριος Καμάλ ε, για τους ε, συντηρητικούς και μεταρρυθμιστές, ο κυρία Βάσκες για τους ΓΚΟΕ και ο κύριος Λάμπερτς για τους πράσινους. Δεν έχουμε για την ώρα σκιώδη από την EFDD. Για, τους, για τα πολυμερή τέλη, τα τέλη των πολυμερών συλλαγών, Ο τριμερής διάλογος συνάρχισε στις 6 Νοεμβρίου. Μπορούμε να αρχίσουμε τώρα τις συζητήσεις. Ε, η ΕΚΟΝ ενέκρινε την ε, συνέχιση του διαλόγου βάσει των αποφάσεων της Ολομέλειας του Απριλίου από τον Ιούλιο. Ο Τριμερής διάλογος λοιπόν θα ξεκινήσει στις 19 Νοεμβρίου το απόγευμα με μια επόμενο γύρο στις 4 Δεκεμβρίου το πρωί. Η διαπραγματευτική ομάδα είναι ο κύριος Ντάλβα Μπιντεγκάιν για το ΕΛΚ, ο κύριος Λούπτιξον για τους σοσιαλιστές, ο κύριος Σαμποτέρο Τέρχο για τους συντηρητικούς και μεταρρυθμιστές, η κυρία Ίντβελτ για τους φιλελεύθερους, ο κύριος ε, Κάφη για την ε, Γκουε και ο κύριος Έκχαουτ για τους πρασίνους μαζί με τον κύριο Βάλλη για τους EFTD. Άλλος τρεμερής διάλογος έλαβε χώρα χθες η οδηγία κατά της νομιμοποίησης εσόδων. Ε, η και, ο, ο δεύτερος και τρίτος γύρος έλαβαν χώρα στις 4 και 5 Νοεμβρίου Βάσει του άρθρου 55 εδώ είμαστε συνεπεύθυνοι με την Οπιτροπή ΛΥΜΠΕ και για τις τεχνικές διατάξεις έχει ανατεθεί διαπραγματευτική εντολή ήδη. Τέλος πάντων ίσως δεν χρειάζεται να σας πω την περίληψη όλων των διαπραγματεύσεων. Έχουν προφανώς συζητηθεί πολλά όπως η διαχείριση, η αποτίμηση κινδύνου, και ούτω καθεξής. Ε, επόμενος τριμές διάλογος θα είναι την 3η 26 Νοεμβρίου. Και εδώ βλέπουμε να υπάρχουν πια βήματα πρόοδου και έχουμε την ελπίδα ότι θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε εγκαίρως αυτό το σημαντικό νομοθέτημα. Να προχωρήσουμε στο τρίτο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Μηνιαία χρονοθυρίδα για τις εξουσιοδότηση πράξεις και τα εκτελεστικά μέτρα και τον έλεγχό τους από τη δική μας πλευρά. Ένα νέο στοιχείο της σημερινής διάταξης που δείχνει την αφοσίωσή μας στο σκοπό μας αυτές οι κατεξοδότηση πράξεις και τα εκτελεστικά μέτρα να ελέγχονται ενδελεχώς και διεξοδικώς και προκειμένου να εκπληρώνουμε τα θεσμικά τις θεσμικές και δημοκρατικές μας αρμοδιότητες. Σήμερα έχουμε τέσσερα θέματα, τις κατεξουσιοδότητες πράξεις και τα εκτελεστικά μέτρα που αφορούν την φεραγγιότητα 2, το Solvency 2, το δίκτυ κάλυψης ρευστότητα για τα χρηματοποστατικά ιδρύματα βάσει του κανονισμού βάσει του κανονισμού για τι κεφαλαίκες απαιτήσει και βάσει του άρθρου 429 καθώς και την υποβολή εκθέσεων αναχώρα σύμφωνα με το άρθρο 89. Και την οδηγία για την ανάκαμψη και την εξυγίανση των πιστοτικών ιδρυμάτων με τον ενιαίο μηχανισμό εξυγίανσης. Η τέταρτη αυτή κατεξοσοδότηση πράξη έχει περισσότερο περίπλοκη θεσμική φύση, διότι αποτελείται από δύο στοιχεία. Την κατεξοσοδότηση αυτή πράξη την, έχουμε, την έχει διεγκρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όμως συμφωνήσαμε να περάσει ως πακέτο. Τα εκτελεστικά λοιπόν μέτρα δεν έχουν εγκριθεί ακόμη. Ούτε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα το κάνει αυτό τις προσεχείς ημέρες προκειμένου να μπορέσει να επιφέρει τροπολογίες και το Συμβούλιο και συμφωνήσαμε με τον Συμβούλιο και ελπίζουμε να συμφωνήσει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφωνήσαμε να υπάρξει μια διαδικασία που θα επιτρέψει την έγκριση και την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων στο Συμβουλίο να τα λάβουμε υπόψη πρωτού αποφασίσουμε για τα εκτελεστικά μέτρα για να δούμε τι θα γίνει και με την κατεξοδότηση πράξη για την οποία έχουμε τη διαδικασία πιθανής αντίρρησης. Ε, θα τα αντιμετωπίσουμε λοιπόν ως πακέτο, ως δέσμια αυτά τα δύο νομοθετήματα και ευχαριστούμε το Συμβούλιο για την προθεμία του να συνεργαστεί μαζί μας. Τους ευχαριστούμε για την καλή τους διάθεση να δουν μαζί μας τα επόμενα βήματα της αξιολόγησης. Και βεβαίως ε, ε, αναμένουμε και την ενημέρωση του Κοινοβουλίου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ως προς αυτά, να πω ότι δεν είμαστε πλήρως ικανοποιημένοι λόγω λόγω της έλλειψης συζήτησης για κάποια σημεία των εκτελεστικών μέτρων, τα οποία δεν είναι απλώς λεπτομέρειες, αλλά έχουν τεράστιο αντίκτυπο στον καταμερισμό των τελών, ε, στον καταμερισμό μάλλον των κονδυλίων, αυτά θεωρούμε ότι δεν έχουν γίνει αντικείμενο ε, σωστής ενημέρωσης προς το Κοινοβούλιο με τους επίσημους διάβλους της θεσμικής ενημέρωσης. Όταν τα έχουμε μάθει είναι από άλλε πηγέ. Ελπίζουμε λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιδείξει πλήρη διάθεση συνεργασία και να ενημερώνει το Κοινοβούλιο για κάθε βήμα πρόοδου ε, στη διαδικασία αυτή και για οποιαδήποτε απόφαση μπορεί να επηρεάζει αυτέ τι αποφάσει, όπου μπορεί να έχουμε και εμεί κάποια θεσμική αρμοδιότητα όπω για τις εξουσιοδότηση πράξη. Ελπίζουμε λοιπόν να βελτιωθεί ο μηχανισμό ανταλλαγή πληροφοριών για τέτοια θέματα. Πρώτο σημείο λοιπόν, φερεγγιότητα 2. Ναι, παρακαλώ για το σημείο αυτό. Για το τελευταίο σημείο έχω μία παράκληση σε ό,τι αφορά την διαδικασία, σε ό,τι αφορά το τελευταίο σημείο. Λοιπόν, ήθελα να το εξή να διευκρινίσω. Νόμιζα ότι θα είχαμε συζήτηση σήμερα. Δεν θα ήθελα μεγάλη συζήτηση, αλλά μία παράκληση από πλευράς, προς την γραμματεία από πλευράς μας να ελέγξουμε κατά πόσον ε, οι παρεκκλήσεις που έχουν ε, κοιτάξει σε ό,τι αφορά το μέγεθος και το κίνδυνο που διατρώχουν οι τράπεζες, κατά πόσον αυτό είναι επιτρεπόμενο ή αν πρόκειται για επίπεδο 2 και αν ξεπερνάμε αυτό που προβλέπει το επίπεδο 1 του PRD. Ο κύριος Χουκμαρκ είπε σωστά ότι το ανώτατο όριο θα πρέπει να είναι το PRD, αλλά θεωρώ ότι αυτό πλέον δεν είναι δεδομένο και, γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα η νομική υπηρεσία να το ελέγξει αυτό. Θα ήμουν πολύ ευγνώμων. Θα επανέλθουμε σε αυτό έτσι και αλλιώς θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο της σας διαταξής. Να πάμε τώρα όμως στο solvency, στη φραγκαιότητα γιατί και οι άλλοι συγκεκριτές θα πρέπει να φύγουν ενδεχομένως. Να δώσω λοιπόν κατευθείαν το λόγο στην κυρία Στέλλερ. Στις 9.30 ε, έχω και τριμερή διάλογο, γι' αυτό θα πρέπει να σπεύσω σε λίγο. Η απόφαση λήφθη το 2009 για τι κατεξόδα τη πράξη. Πρώτη συνεδρία των σχεδόν τον έγινε στο περασμένο Στρασβούργο για να δούμε τι αρχικέ απόψει των ομάδων. Η πράσινη είναι κατά των κατεξοδότηση πράξεων και φαντάζομαι θα μας εξηγήσει ο εκπρόσωπος τους, ο συντονιστής τους, τους λόγους για την απόρριψη αυτή. Ε, έχουμε συνάντηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σήμερα και την επόμενη εβδομάδα με την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων, την ΕΙΟΠΑ. Και φυσικά προσβλέπουμε στην έναρξη των τεχνικών συζητήσεων, γιατί έχουμε κάποιε εκκρεμότητε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ΕΙΟΠΑ, την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων. Λυπούμε, αλλά πρέπει να φύγω, όπω σα είπα, έχω τριμερή διάλογο θα πρέπει να σας εγκαταλείψω. Ευχαριστώ πάντως προβλέπω στις συζητήσεις και ευχαριστώ τη Γραμματεία για το έργο της. Πάντως η 12η Ιανουαρίου είναι η ιανουαριου ειναι προθεσμία για την υποβολή αντιρρήσεων. Οπότε αν δεν υποβληθούν αντιρρήσεις ή στάσεις, θα αρχίσουμε από την 1η Απριλίου του επόμενου έτους. Thank you. Now the first... Ευχαριστούμε. Πρώτο σκιώδης, ο κ. Πάλις από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς ε, να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη σημερινή ανταλλαγή απόψεων. Έχουμε πλέον ε, τις, ε, τα σχέδια για τις πράξεις κατεξιοδότηση για το Solvency 2. Εμείς θα θέλαμε να έχουν κατατεθεί πιο νωρίς βέβαια, μέσα Οκτωβρίου. αυτές οι πράξεις κατά εξουσιοδότηση θα πρέπει να φροντίσουν ε, να υπάρχει συνέπεια με την ε, οδηγία. Αυτό που είναι σημαντικό και το επαναλαμβάνω αυτό διαρκώς είναι η αρχή της αναλογικότητας η οποία ενισχύεται στην ε, οδηγία και θα πρέπει να εφαρμοστεί και στις νομοθετικές πράξεις. Και γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να καλήσω εκ νέου την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κοιτάξει ακόμα πιο έντονα θέματα αναλογικότητας ό,τι αφορά τεχνικά στάνταρ, τα τεχνικά πρότυπα και σε ό,τι αφορά την αναφορά αυτή στην αναλογικότητα. Ένα άλλο θέμα είναι οι μακροπρόθεσμες επενδύσεις, ιδιαίτερα στο θέμα των, των υποδομών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, υποχρεώθηκε να κάνει αναθεώρηση μέχρι τα τέλη του 2018. Εμείς θα θέλαμε ήδη τώρα να ε, καλέσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει μια πρόομη αναθεώρηση, γιατί κοιτώντα το πολιτικό περιβάλλον θα πρέπει να θέσουμε και τις ε, ε, απαιτήσει μας. Είναι, νομίζω, σίγουρα δικαιολογημένη μια τέτοια αναθεώρηση. Επίσης, περαιτέρω θα πρέπει να βελτιώσουμε το επενδυτικό κλίμα στην Ευρώπη. Η ασφαλίσεις εδώ νομίζω ότι θα πρέπει να παίξουν σημαντικό ρόλο και θα πρέπει να ληφθούν υπόψη ε, τα θέματα της διαφοροποίησης κινδύνου προκειμένου οι μακροπρόθεσμες ε, επενδύσεις να είναι δυνατές για την πρόθεση της οικονομίας μας. Επίσης θα πρέπει να είναι σημαντικό ότι μπορούμε να κινηθούμε προς τις ε, οδικές, στους αυτοκινητοδρόμους σε ό,τι αφορά τις μακρισμένες περιοχές. Και θα πρέπει να τα λάβουμε όλα αυτά υπόψη. Σε ό,τι αφορά τη συζήτηση για τις επενδύσεις, για την υποδομή με την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με την ΑΙΟΠΑ, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντική και ίσως ε, θα πρέπει να σκεφτούμε κάποια επιπρόσθετα άσθετη. Ίσως η ΑΕΟΠΑ θα μπορούσε να κάνει κάποια τέτοια πρόταση προς την κατεύθυνση αυτή. Κάποια εξημών ήδη στην προηγούμενη θετία και στην προηγούμενη θετία μάλιστα στο... συμμετείχα στην διαδικασία για το Solvency 2. Είχαμε λοιπόν ε, εξαρτητικές συζητήσεις για το Solvency 2. Εγώ το μόνο που έχω να πω είναι ότι πλέον πρέπει να πραγματοποιηθεί και από 1η Ιανουαρίου 2016 να τεθεί σε εφαρμογή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος. Και τώρα για την ομάδα των συντηρητικών και των αριθμιστών, ο κύριος Καμάλ δεν είναι εδώ. Παίρνει το λόγο για το ECR. Α, η Ashley Fox. Αλλά και πάλι. Κανείς. Δεν την βλέπω. Να περάσουμε λοιπόν στην Άλντε. Από την Άλτε. ποιος θα πάρει το λόγο. Κανείς. Από την ΚΟΕ. Ο κύριος Βιέγκας. Ευχαριστώ. για το πακέτο Solvency 2, τα 2, που θέλει ε, κατά βάση να δημιουργήσει μια εναρμονισμένη αγορά στις ασφαλιστικές εταιρείες. Έχω ένα προβληματισμό για τα συνταξιοδοτικά ταμεία. Για το τεχνικό θέμα είναι περίπλοκο και πολύ σύνθετο και χρειάζεται τεχνογνωσία, αλλά έχουμε μια σοβαρή ανησυχία για τον κίνδυνο που ελοχεύει να δώσουμε έμφαση στα καθεστώτα κεφαλαιοποίησης στο συνταξιδοτικό ταμείο εις βάρος ε, των συστημάτων των δημόσιων που στηρίζεται στην αλληλεγγύη. Οπότε το θέμα των ασφαλιστικών εταιριών ε, και των ε, καταστροφών που είχαμε στο Ηνωμένο Βασίλειο γιατί άνθρωποι που έμειναν χωρίς οικονομίες τους εξαιτία ε, χρεοκοπίας ε, συνταξιοδοτικών ε, ταμείων. Αυτό θα πρέπει να το αποφύγουμε. Αλλά κατά τη γνώμη κάθε φορά που συζητούμε το θέμα αυτό, ανακύπτει η βασική αυτή ανησυχία. Πώς θα διαφυλάξουμε κάποια δημόσια συστήματα κοινωνικής ασφάλισης. Και θα πρέπει να δώσουμε σε αυτό το σημείο έμφαση για να προστατεύσουμε και να εξασφαλίσουμε τους εργαζόμενους στα συνταξιδοτικά ταμεία, αν θέλουμε να τα ευνοήσουμε με κάποιους αναδυναμητικούς πυλώνες, αυτά τα στοιχεία θα πρέπει να τα εξετάσουμε, αλλά γενικώ δημιουργούν ένα σοβαρό προβληματισμό και ανησυχία. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε ο κύριος Γκίγκολ για τους πρασινούς. Είχαμε εκτενή συζήτηση για το Solvency 2 και για τα εφαρμοστικά μέτρα. Η κύρια μεταβολή από τις προηγούμενες συζητήσεις. Η κύρια μεταβολή λοιπόν που επηρέασε και τις τελευταίες διαπραγματεύσεις έγκυται στο πώς ε, θα αντιμετωπίσουμε ε, προϊόντα που καλύπτονται από εγγυήσεις. Και να σας ε, πω με δυο λόγια το ιστορικό. Για τέτοια προϊόντα, τριπλού β, ο παράγων κίνδυνος υπολογίστηκε αρχικά τον Οκτώβριο του 2011 και ήταν 20% αυτός ο παράγοντας κινδύνου η ΕΙΟΠΑ ανέλαβε να εξετάσει εις βάθος ε, την ακρίβεια αυτού του υπολογισμού. Για τέτοια προϊόντα υψηλής ποιότητας, τέτοια, ε, διαφορά θα μπορούσε να φτάσει στο 70% για το τρίπλο Β. Μετά η Γενική Διεύθυνση Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής άσκησε πίεση στη Γενική Διεύθυνση για την αγορά και, και μειώθηκε κατά 8,5% στο σχέδιο του Μαρτίου του 2014. Μετά ασκήθηκε ακόμη περισσότερη πίεση και τον Ιούλιο του 2014 μειώθηκε από το 8,5% στο 5%. Τώρα ο παράγοντας, ε, το ποσοστό που βλέπουμε και μας προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, μειώθηκε ακόμη περισσότερο, 3%. Τι γίνεται για τα προϊόντα με 3α, διπλό α ε, και α. Τι σημαίνει. Σημαίνει ότι ο παράγοντας κινδύνου των προϊόντων δεν εξαρτάται από εμπειρικές αποδείξεις των χρηματοπιστωτικών αγορών, αλλά επηρεάζεται από πολιτικούς στόχους. Και αυτό ήδη ισχύει στον κανονισμό για τις τράπεζες και τις ασφάλισεις ό,τι αφορά τα κυβερνητικά ομόλογα. Εκεί, στην περίπτωση των κυβερνητικών ομολόγων, των κρατικών ομολόγων, οι χώρες ε, προσπαθούν να διαβεβαιώσουν τους ε, ενδιαφερόμενους ότι δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος και τώρα δημιουργούμε μια δεύτερη κατηγορία στοιχείων του ενεργητικού, τα εξασφαλισμένα προϊόντα που λένε ότι ο κίνδυνος είναι πολύ λιγότερος από ό,τι θεωρεί η αγορά. Αυτά τα τιτλοποιημένα προϊόντα. Ενώ και προσπαθούμε να πείσουμε τις αγορές ότι η κατάσταση είναι πέντε φορές καλύτερη από ό,τι στην ουσία είναι. Αυτό κάνει το κράτος, αλλά το κράτος κανονικά θα πρέπει να ρυθμίζει τις ασφαλίσει και τι ασφαλιστικέ εταιρείε, ώστε να έχουν οι εταιρείε αρκετό κεφάλαιο για να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσει του. Οπότε είναι σημαντικό η μελέτη του κινδύνου, η αξιολόγηση του κινδύνου, να λαμβάνει και κάποια κριτήρια προφύλαξη. Εδώ προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε χρηματοπιστωτικό κανονισμό προκειμένου να τονώσουμε την οικονομική ανάπτυξη. Συμφωνώ με τον κύριο Μπάλτς ότι οι ασφαλίσεις είναι σημαντικός κλάδος για τις επενδύσεις. Αλλά δεν δικαιολογείται αυτή η σημασία από την πολιτική επέβαση και ε, τον πολιτικό επηρεασμό ή την πολιτική παρουσίαση ή μείωση τεχνικά του παράγοντα κινδύνου. Γιατί μια τέτοια δραματική μείωση του κινδύνου θα πρέπει να δικαιολογείται. Γιατί μειώσατε τόσο δραστικά τα ποσοστά αυτά παρά τις, τα επιστημονικά πορίσματα που κατέθεσε η ΕΙΟΠΑ μετά από τεκμηριωμένη και δελεχή μελέτη. Ακριβώς για να τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμα ζητήσαμε να γίνει ψηφοφορία και αύριο θα έχουμε συνεδρίαση την οποία ζητούσαμε εδώ και πολύ καιρό και αύριο θα συζητήσουμε το θέμα αυτό με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ελπίζω να είναι εκεί και εκπρόσωπος της ΕΙΟΠΑ. Πάντως σας προειδοποιώ θα κάνουμε το ίδιο λάθος με τις Ηνωμένε Πολιτείε. Ουσιαστικά εθελοτυφλούμε στο κίνδυνο που υπάρχει και κάποια ενυπόθηκα προϊόντα δεν ε, υποχρεώνουν τους ενδιαφερόμενους να έχουν επαρκές κεφάλαιο γιατί αυτό που μας ενδιαφέρει υποτίθεται είναι μόνο η οικονομική ανάπτυξη. Μας ενδιαφέρει και η οικονομική ανάπτυξη και σίγουρα η αηφόρος ανάπτυξη αλλά δεν θα πρέπει η χρηματοπιστωτική ρύθμιση, ο χρηματοπιστωτικός κανονισμός ε, να αναλαμβάνει αυτό το ρόλο. Δεν θέλουμε μία ε, κατηγορία, δεύτερη κατηγορία στοιχείων του ενεργητικού, όπου το κράτος θα γνωρίζει καλύτερα ποιος είναι ποιο είναι το ποσοστό του κινδύνου. Θα πρέπει να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτά τα τιτλοποιημένα προϊόντα. Και νομίζω ότι την ίδια συζήτηση θα έχουμε όταν θα μιλήσουμε για το LCR, το δίκτυο κάλυψη ρευστότητα. Περιμένω διεξοδικέ εξηγήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα στηρίζεται σε πραγματικέ αποδείξει και θα μα τεκμηριώσει το χαμηλό ποσοστό κινδύνου που προτείνει. Ευχαριστώ. Πριν δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να δώσω το λόγο στην κυρία Ελίζα Φερέιρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να Ζήτησα το λόγο όχι για να περάσω σε σχόλια για το περιεχόμενο όπως άλλοι συνάδελφοι, αλλά να επιστήσω την προσοχή της Επιτροπής στην ανάγκη να προσκαλέσουμε την ΕΙΟΠΑ να ερευνήσει και να δουλέψει στο πώς πρέπει για τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις να προβλέψουμε μια άλλη κατηγορία στοιχείων του ενεργητικού, διότι η κατηγορία αυτή ε, είναι ένα αντιστάθμισμα για τις ε, μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις που ε, είναι επίσης και η βάση για τις ασφάλειες. Χρειαζόμαστε λοιπόν μια κατηγορία στοιχείων του ενεργητικού με μεγάλη διάρκεια και θα πρέπει να κληθεί η ΟΠΑ από εμάς με πολύ μεγάλη σαφήνεια να προτείνει μια κατηγοριοποίηση, μια στάθμιση των ε, σχετικών προϊόντων βάσει του Solvency 2 και αυτή η κατηγορία να χρησιμοποιηθεί ώστε μακροπρόθεσμα να υπάρχουν βιώσιμες επενδύσεις και οι ανάλογοι στόχοι από την Ευρώπη. Αυτό το μήνυμα ήθελα να αποστείλω και εφόσον υπάρχει συμφωνία μεταξύ των πολιτικών ομάδων, παρακαλώ να προωθήσουμε το αίτημα αυτό προς την ΕΟΠΑ. Σας ευχαριστώ και τώρα από το ΕΛΚ, αν σωστά κατάλαβα, ε, διατυπώθηκε ένα παρόμοιο σχόλιο. Άρα υπάρχει ήδη μια κάποια πλειοψηφία για την πρόταση αυτή. Τώρα κανένα άλλο συνάδελφο θέλει το λόγο. Ωραία. Άρα να δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριος Κλάους Βίτνερ. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Ναι, δύο-τρεις γενικές παρατηρήσεις και θα προσπαθήσω να απαντήσω στις ερωτήσεις που ακούσαμε σήμερα το πρωί για το Solvency 2. Όλοι θα ξέρετε ότι το έχουμε εδώ και πολύ καιρό. Αντικαθιστά 40 ε, ήδη φυστάμινε οδηγίες. Θα είναι πρώτος τέτοιος ενιαίος κανόνας και θα υπάρχει μια ενιαία ευρωπαϊκή προσέγγιση πλέον σε ό,τι αφορά τις ε, απαιτήσει ω προ την αξιολόγηση κινδύνου. Πρόκειται για ένα από τα πιο προηγμένα παγκόσμια συστήματα και αυτό το αναγνωρίζουν και άλλε χώρε, τρίτε χώρε, οι οποίε αλλάζουν πλέον και προσπαθούν να προσεγγίσουν το Solvency 2. Νομίζω ότι αυτό είναι το καλύτερο κοπλιμέντο που μπορούμε να έχουμε. Αυτό θα πρέπει να είναι το σημείο κίνηση. Το σημείο αφετηρία. Έχουμε πλέον το τελευταίο βήμα τη πράξη κατά εξουσιοδότηση ουσιαστικά. Προφανώ και είναι σημαντικό. Και όλοι συμφωνούμε ότι οι πράξει κατά αξιοδότηση θα πρέπει να συμμορφώνονται με το επίπεδο 1. Προσπαθήσαμε να είμαστε όσο πιο ανοιχτοί και όσο πιο διαφανεί μπορούσαμε. Προφανώ έγιναν και πάρα πολλέ ε, συναντήσει από το 2009 με του εμπειρογνώμονες των κρατών μελών, με τι γραμματείε, πολλέ ε, άτυπε επαφέ, ε, με τα κράτη-μέλη, επίσημε επιστολέ. Όλα αυτά ελήφθησαν υπόψη όσο πιο διαφανείς μπορούσαμε είμαστε. Και σε τελική ανάλυση θεωρώ ότι το κείμενο α, είναι του καλύτερου δυνατόν από πλευράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παρούσα χρονική συγκυρία. Για να επισέλθουμε τώρα στα δύο βασικά θέματα. Οι μακροπρόθεσμες επενδύσεις προφανώς και αποτελούν έναν σημαντικό στόχο. Αλλά όχι εις βάρος της προστασίας των ε, ναι, πολιτικών αυτών. Και γι' αυτό λοιπόν στην παρούσα φάση δεν συμπεριλάβαμε την υποδομή, γιατί δεν μας ικανοποιούσαν τα δεδομένα που είχαμε για τον ορισμό της υποδομής, των υποδομών, για να συμπεριληφθεί, για να δημιουργηθεί μια ξεχωριστή κατηγορία. Προφανώς είμαστε ανεκτοί για να δημιουργηθεί μια τέτοια κατηγορία το συντομότερο δυνατόν και να αλλάξουν μετά οι πράξει κατά εξουσιοδότηση. Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι στην παρούσα φάση το Solvency 2 μέχρι το 2016 είναι σημαντικό και στο παγκόσμιο προσκήνιο και στις επιχειρήσεις γιατί όλες έχουν προετοιμαστεί και τώρα λοιπόν πρέπει να έχουν επιτέλους τις ημερομηνίες, τις προθεσμίες. Θα ήταν λοιπόν σπατάλη πόρων να αλλάξει η προθεσμία. Αναθεώρηση, εντάξει, να το κοιτάξουμε, να προσπαθήσουμε να το προσαρμόσουμε κατά το δυνατόν, αλλά να μείνει η ημερομηνία 1η Πρώτη του 2016 σε ό,τι αφορά την τιτλοποίηση. Όντω, κοιτώντα τα θέματα τιτλοποίηση, νομίζω ότι είναι ένα τεράστιο βήμα ότι για πρώτη φορά στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία έχουμε τον ορισμό τη υψηλή ποιότητα τηλεοποίηση μαζί με τι πράξει κατοξιοδότηση για το ΕΣΥΑΡ, το οποίο θα συζητήσουμε σε λίγο. Το πρόβλημα ήταν στο παρελθόν ότι η τυκλοποίηση ήταν απλά τυκλοποίηση και αυτό ήταν λάθος, γιατί δεν ξέραμε τι σήμαινε ακριβώς, δεν υπήρχε διαφάνεια. Αυτός που είχε κάνει τη τιτλοποίηση δεν, έκανε, δεν διατρέχει κίνδυνο και προφανώς αυτό ήταν μία από τις αιτίες που οδήγησαν στην κρίση. Γι' αυτό λοιπόν ήταν τόσο σημαντικό σε αυτό το κείμενο να υπάρχει σαφή να υπάρχουν σαφή κριτηρία για την υψηλή ποιότητα λειτουργοποίηση. Θα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια, θα πρέπει να υπάρχει ομογένεια. Όλα αυτά είναι κριτήρια τα οποία διασφαλίζουν ότι δεν θα αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα των περασμένων ετών. Και εκ παραλλήλου πρέπει να έχουμε υπόψη ότι θα πρέπει να προσθέσουμε κάτι που θα συνάδει με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Να υπάρχει δυναμικό ασφαλές και το οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε χωρίς να βλάψουμε την πολιτική για την προστασία. Δύο πράγματα θα πρέπει να λάβουμε υπόψη σε σχέση με την κρίση. Έχουμε, έχετε αλλάξει την νομοθεσία πλέον και έχει ξεκαθαριστεί ότι πλέον υπάρχει περιορισμός κινδύνου. Δεν λαμβάνουμε υπόψη Λοιπόν, ε, πρέπει να πάρουμε υπόψη και τον κίνδυνο και να περιορίσουμε κάποιον τον κίνδυνο τη και παράλληλα έχουμε και τις ε, εποπτικούς ε, οργανισμούς. Αυτά λοιπόν από κοινού μας δίνουν τη δυνατότητα να έχουμε την αξιολόγηση που προτείνουμε. Το πρόβλημα με την τηλεοποίηση δεδομένων ήταν ότι τα δεδομένα που είχε η ΟΠΑ ήταν τα δεδομένα της κρίσης, των ετών της κρίσης. Προφανώς αυτό ήταν απαραίτητο αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τις αλλαγές που έχουν γίνει. Και το γεγονός ότι προφανώς ένας από τους βασικούς λόγους για την αξιολόγηση που έχουμε τώρα είναι αυτό που ονομάζουμε look-through. Το οικονομικό επιχείρημα είναι ότι όταν ενώνουμε, συνενώνουμε δάνεια, διαφοροποιούμε τον κίνδυνο. Και αυτές που είναι πιο ασφαλείς, είναι δύσκολο να πούμε ότι ακόμα και αυτές θα ήταν πιο επικίνδυνες από τα αν παίρναμε ένα μόνο δάνειο ξεχωριστά. Αυτό είναι οικονομικό επιχείρημα και το οποίο έχει δοκιμαστεί. Και νομίζω ότι στέκει ακόμα. Αυτό λοιπόν ε, θα πρέπει να περιοριστεί. Σας ευχαριστώ πολύ. Yes, ε, Πολύ γρήγορα. Ε, με συγχωρείτε αλλά νομίζω δεν απαντήσατε στην ερώτησή μου. Προασπιστήκατε τον ορισμό για την υψηλή ποιότητα στην κλοποίηση, αλλά δεν σας είπα εγώ ότι αυτό με ενοχλεί. Δεν ε, είμαι κατά της υψηλής ποιότητας ε, τα τυπλοποιημένα προϊόντα, αλλά έχουν συγκεκριμένο οικονομικό ρόλο να διαδραματίσουν. Και ρώτησα συγκεκριμένα ποια είναι τα στοιχεία σας, τα πρακτικά στοιχεία, για να μειώσετε κατά πέντε την στάθμιση του παράγοντα κινδύνου. Μπορείτε να μας παρουσιάσετε πρακτικά στοιχεία, ε, δεδομένα που να το στηρίζουν αυτό, να στηρίζουν αυτή την αλλαγή. Εάν υπάρχουν, καλό θα ήταν να καταλάβουμε πώς ε, φτάσατε σε αυτόν τον αριθμό, ενώ εμείς έχουμε στοιχεία από την πράξη, από την ΕΟΠΑ από τον Ιανουάριο του 2014, που αποδεικνύουν το αντίθετο. Επιτροπή θέλετε να απαντήσετε. Ναι, ήδη έχω δώσει κάποια στοιχεία απάντηση. Η ΟΠΑ πήρε τα στοιχεία από την περίοδο της κρίσης, αλλά αν συγκρίνεται τι συνέβη με άλλα νομοθετικά, με άλλα μέσα, με άλλα εργαλεία μάλλον, όπως τα καλυμμένα ομόλογα, βλέπετε ότι ελάζει ο παράγοντας κινδύνου αν πάει κανείς πίσω από την προηγούμενη πενταετία. Αυτό δείχνει ότι τα δεδομένα δεν αρκούν για να έχουμε μια συνολική εικόνα. Αυτό ήταν ε, το πρώτο στοιχείο. Το δεύτερο είναι ότι η ΟΠΑ χρησιμοποίησε δεδομένα, δεδομένα κρίσης τη στιγμή που δεν είχαμε τον κανονισμό που έχουμε τώρα. Τι σημαίνει αυτό. Ισχυάν άλλοι κανόνες. Είχαμε τους ε, οργανισμούς ε, αξιολογίας που δεν τους επιβλέπει η ΕΣΜΑ ένα σωρό διαφορές που τώρα πρέπει να λυθούν υπόψη. Η ΕΟΠΑ πήρε τα δεδομένα, αλλά δεν είδε τη συνολική εικόνα. Και όπως είπα, το πλέον σημαντικό επιχείρημα που τελικά μας έπεισε κιόλα είναι το look-through. Πώς να πείσουμε κάποιον ότι αν διαφοροποιηθεί ο κίνδυνο και αν πάρουμε μόνο τα μερίδια σύνορα αυτών που δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση να πτωχεύσουν, δεν είναι πιο επικίνδυνο από το να πάρει κανεί ένα μόνο δάνειο από κάποιον που δεν έχει, σαφή που έχει ένα συγκεκριμένο παράγοντα κινδύνου. Έτσι, έτσι χρησιμοποιήσαμε το επιχείρημα του δάνειο. δανείου. Με συγχωρείτε, δεν μου απαντάτε, δεν μου απαντάτε ποια είναι τα δεδομένα σας. Φυσικά, εάν το βγάλετε εκτός, από τη, εκτός χρονικού πλαισίου τα χρόνια της κρίσης, φυσικά είναι πιο συμπαθητικά τα δεδομένα. Όμως, τα δικά σας δεδομένα που είναι, ποια είναι η λογική σας βάση για το 5% στο τριπλό β. Ε, κοιτάξτε το από μια άλλη οπτική γωνία. Υπάρχει μια στάθμιση για τα δάνεια 3%. Το ερώτημα είναι, εάν τιτλοποιηθούν τα δάνεια αυτά, και πάρει κανείς μόνο τα senior ε, σκέλη τους. Θα πρέπει να γίνει πιο ε, υψηλή, σε, υψηλότερη κατηγορία η στάθμιση. Μα κοιτάξτε αν λένε οι οίκοι ότι είναι τριπλό δίτα. και εσείς λέτε 20% στα χρόνια της κρίσης και το μειώνετε στο 3% και κατά της αξιολόγησης κινδύνου από, τα, από τους οίκους ε, αξιολόγησης. Ε, πού είναι η συμφωνία. Με συγχωρείτε, αλλά εγώ αυτό που ήθελα να καταλάβω το κατάλαβα. Δεδομένα δεν υπάρχουν. Επιτροπή θα προσθέσετε κάτι. Ε, κοιτάξτε, εδώ δεν παίζουμε το ρόλο των οίκων αυτό που κοιτάζουμε είναι τι συμβαίνει στο ε, βασικό δάνειο. Εκεί, αν αποδεχτείτε το 3% πρέπει να αποδεχτείτε και τα σκέλη που είναι senior ε, και, τις δύο, και στις δύο περιπτώσεις. Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι και οι δύο θέσεις είναι πολύ σαφείς. Οπότε μπορούμε να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση για το θέμα αυτό και να θυμίσω ότι σε ό,τι μας εφόσον λάβουμε πρόταση από τους πρασίνους, θα ξεκινήσει η εσωτερική διαδικασία υποβολής αντίρρησης που μπορεί να λάβει χώρα θεωρητικά στην Σύνοπελομέλειας του Δεκεμβρίου, εφόσον υπάρξει πλειοψηφία, κάτι που δεν διαφαίνεται από αυτή τη συζήτηση, αλλά η διαδικασία πρέπει να ακολουθηθεί. Και αυτό θα γίνει. Επίσης, να πω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι σημειώνω αυτά που είπατε και αυτά που σημείωσαν δύο ε, πολιτικές ομάδες για την περισσότερο διερεύνηση και έρευνα της ε, δομής της κατηγορίας των μακροπρόθεσμων στοιχείων του ενεργητικού. Δεν κατάλαβα εάν συμφωνήσατε ότι να ζητήσουμε εμείς από την ΕΟΠΑ να αρχίσει να το μελετά αυτό. Επιτροπή. Νομίζω ήδη έχουν προθυμοποιηθεί να το αντιμετωπίσουν το όλο θέμα και εμεί του ενθαρρύναμε. Οπότε ναι, μπορείτε να συνεχίσετε. Πρόεδρο, ευχαριστούμε. Περνάμε λοιπόν στο δεύτερο σημείο που είναι ο δείκτη κάλυψη ρευστότητα και ο δείκτη μόχλευση. Θα ήθελα ευθύ αμέσω να δώσω το λόγο, εφόσον έχει εγκριθεί αυτή η κατεξοσοδότηση πράξη από τον Οκτώβριο, θα ήθελα να δώσω ευθύ αμέσω το λόγο στον εισηγητή που είναι ο κύριος Ατμαρκάρας. Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι αγαπητοί συνάδελφοι, θα ξεκινήσω με το θέμα του α, ποσοστού χρέωσης, γιατί είναι πιο απλό. Από δική μου πλευράς δεν υπάρχουν άμεσες αντιρρήσεις, αλλά μία ερώτηση επί του περιεχομένου. Τα πρότυπα για το reporting, για την αναφορά για το έτος 2015 γιατί ήδη για την ΕΠΑ. Από την ΕΠΑ. Αυτό που άκουσα σε πολλές περιπτώσεις είναι ότι υπάρχει ανασφάλεια, αβεβαιότητα ε, βάσει ποιων templates, ποιων προτύπων θα γίνει η δηλώσει, η αναφορά για το πρώτο τετράμινο, τρίμηνο. Γιατί δεν είναι σαφές. Ερωτώ λοιπόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχει κάνει συζητήσεις με την ΕΠΑ εδώ για το πότε θα δημοσιευθούν αυτά τα νέα, είναι οι πίνακες, τα νέα πρότυπα αυτά. Ή υπάρχει από πλευρά σας και σκέψεις ε, για την πρώτη αναφορά το 2015, μήπως χρησιμοποιηθούν τα παλιά πρότυπα, τα παλιά templates, οι παλιοί πίνακες. Δεύτερο θέμα, πολύ πιο δύσκολο. Ελάχιστο ποσοστό ρευστότητας. Χαίρομαι που υπάρχει επιτέλους ε, σαφήνεια για το πώς ε, μπορούν να πετύχουν τα ιδρύματα την απαραίτητη ρευστότητα, αλλά σε ακριβή ανάλυση των δύο κειμένων για το End Level 2 βλέπουμε ότι συναντάμε κάποια προβλήματα όπου χρειαζόμαστε διευκρινήσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κατά πρώτον, γιατί υπάρχει διαφορετικός ορισμός των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο level 1, στο πρώτο επίπεδο 1 και στο υπόλοιπο. Δεύτερο, και σε ό,τι αφορά τους ιδιωτικούς πελάτες, τους ιδιώτες. Υπάρχουν διαφορές στα νομικά κείμενα. Στο σύρα. υπάρχει δεσμευτικότητα και δέσμευση για, για φυσικά πρόσωπα και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Στο ε, κείμενο του επίπεδου 2 μόνο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δηλαδή, συνειδητά εξαιρούμε εδώ τα φυσικά πρόσωπα ή κατά λάθο έγινε αυτό. Τρίτον, στην τελευταία πρόταση του 418.4 αναφέρεται στο CR ότι η ορθότητα ενός υπολογισμού θα πρέπει να ελεγχθεί από εξωτερικό ελεγκτή. Στην πράξη καταξουσιοδότηση αυτό το απόσπασμα δεν εμφανίζεται πλέον. Άρα οι τράπεζες ποιο νομικό κείμενο πρέπει να επικαλεστούν. Υπήρξε μείωση το μηχανισμό ε, ελέγχου των τραπεζών που μπήκε από παραθυράκι γιατί κάθε μείωση ελέγχου δεν θα εγκριθεί από το Κοινοβούλιο. Τέταρτον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι σκέφτεται σε ό,τι αφορά τις τρεις διαφορές των κειμένων. Χρειάζεται διευκρίνηση, χρειάζεται διορθωτικό από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Προβλέπετε τι νομοθετικά κείμενα θα χρησιμοποιήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε ό,τι αφορά τη διάκριση μεταξύ επίπεδου 1 και 2. Εμείς δεν θα επιτρέψουμε υπονόμευση του νομοθέτη μέσω της πίσω πόρτας. Γι' αυτό λοιπόν κάθε αντίφαση θα πρέπει να διευκρινιστεί. Thank you. Σας ευχαριστώ. Και τώρα θα δώσω το λόγο στους σκιώδη ηγητές. Πρώτα στον ε, σκιώδη ηγητή των Σοσιαλιστών Δημοκρατών, στον κύριο Ούντο Μπούλμαν. Ε, θα ήθελα να συγχαρώ τον Ότμαρ καταρχήν για τη σωστή αξιολόγηση και την αξιόλογη προσπάθεια που έκανε για αυτό το τμήμα της καταξιοδότησης πράξης και περιμένω με ανυπομονησία την απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εκπρόσωπος των συντηρητικών μεταρρυθμιστών, δεν βλέπω τον Καμάλ εδώ. Άλλος κανείς από την ΙΣΙΑΡ για να αντικαταστήσει τον Καμάλ Μιχαήλ Τόιερ. Θα θέλετε το λόγο για τους φιλελεύθερους. Δεν ανάβετε το μικρόφωνο για να σας ακούμε κι εμείς. Ε, δείκτης κάλυψη ρευστότητας το θέμα μας. Από την ΚΟΥ ο κύριος Βιέγκας. Εγώ προβληματίζομαι κάπως γιατί προέρχομαι από ακαδημαϊκούς κύκλους και από θέματα οικονομίας και άλλα λέμε στους ε, φοιτητές μας και άλλα ακούμε εδώ. Γιατί προσπαθούμε εδώ να ρυθμίσουμε μια πραγματικότητα που είναι απείρως πολυσύνθετη. Ο κόσμος είναι περίπλοκος και πολύπλευρος. Εδώ θέλουμε να περιχαρακώσουμε τον, τον κίνδυνο και τη ρευστότητα ενώ έχουμε πολύ περίπλοκους παράγοντες που είναι αδύνατο να πραγματικά να τους λάβουμε υπόψη. Οπότε Κατά ανάγκη γινόμαστε κάπως πιο αυθαίρετοι στους ε, δείκτες, ε, στους λόγους, στη στάθμιση των στοιχείων του ενεργητικού. Στο σενάριο των ροών, των νομισματικών των ε, ροών που καθορίζουν το δίκτυ κάλυψης ρευστότητας. Προσπαθούμε στην ουσία να ρυθμίσουμε μια πραγματικότητα που είναι πολύ πιο πολυσύθετη και περίπλοκη. Αυτή η προσπάθεια ενέχει κινδύνους που τους βιώσαμε και στο παρελθόν. Γιατί πολλές φορές η νομοθεσία μας δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, γιατί δεν μπορεί να συλλάβει την πραγματικότητα στην περιπλοκότητά της. Και ε, απαιτεί και από την αγορά να προσαρμοστεί και πολλές φορές να παρακάμψετε τους κανονισμούς. Για το, το λόγο κάλυψης ρευστότητας ακούσαμε πολλές επικρίσεις και την πιθανότητα κάποιων φορέων, ακριβώς επειδή μπορούν να, να τηρήσουν αυτούς τους λόγους κάλυψης ρευστότητας, να επικεντρωθούν υπερβολικά σε βραχυπρόθεσμες ενέργειες. Επίσης έχουμε συμπεριφορές από τράπεζες, από φορολογικούς παραδείσους που μας δημιουργούν πολλές αμφιβολίες για την αποτελεσματικότητα μιας τέτοιας νομοθετικής ρύθμισης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κάποιος από τους πρασίνους. Σβέν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ τον Ότμαρ Κάρας για την εμπεριστατωμένη ανάλυση που μας έκανε. Έχω μία ερώτηση. Τι θεωρεί η ή ο κανονισμός. Το άρθρο 416 παράγραφος 2. Ότι μόνο τέτοια προϊόντα θα πρέπει να θεωρούνται ως υψηλής ρευστότητας αν αποδειχθεί ότι έχουν την, δυνα... την καλύτερη δυνατή ποιότητα της Ευρωπαϊ... Ε, όπως κρίνει η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών θα κρίνει ποια προϊόντα είναι ποιοτικά. Ενώ στην έκθεσή τους, στην έκθεση της Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών που έπρεπε να υποβάλει στα τέλη του 2013 δεν θεώρησε ότι τα καλυμμένα ομόλογα ή τα δάνεια SME ή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ή τα καταναλωτικά δάνεια ενέπιπταν σε τέτοια στοιχεία του ενεργητικού και δεν υπήρχε κάτι τέτοιο στις ε, ε, συστάσεις της ε, Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, αλλά και πάλι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φαίνεται να θεωρεί ότι ξέρει καλύτερα τα πράγματα. Μήπως έτσι όμως παραβιάζει τον κανονισμό. Και δεύτερον, γιατί ε, όπως πρόβλεπε η νομοθεσία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ακολούθησε τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών. Επίσης πληρούνται εδώ οι διατάξεις της Βασιλείας γιατί η τρίτη τη ρυθμίση της Βασιλείας ε, είπε να περιοριστεί σε κρατικά ε, σε δημόσιο χρέος. Δεν αναφέρονται ούτε τα ε, καλυμμένα δάνεια, ούτε τα ABS. Οι τίτλοι προερχόμενοι από τιτλοποίηση δηλαδή. Τι θεωρεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τη γνωρίζει καλύτερα από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών ή τη Βασιλεία. η τη βασιλεια Ευχαριστώ για το EFTD. Κανείς δεν είναι εδώ, εντάξει. Δεν έχουμε και κάτι στη DI. Θα δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο κύριο Νιάν Μπόγαν. Good morning thank you for... Καλημέρα σας και ευχαριστώ για την ευκαιρία να σας απαντήσω στις ερωτήσεις. Να ξεκινήσω με την ερώτηση για, το, για τη συλλογιστική αυτή τη κατεξοδότηση πράξη. Να θυμίσω ότι η κρίση έδειξε ότι υπάρχουν κάποια κενά και ελλείψεις στο νομοθετικό μας πλαίσιο. Το single book, το ενιαίο εγχειρίδιο κανόνων για τις τράπεζες, είχε πολλές ελλείψεις και είδαμε ιδίως στον τομέα της ρευστότητας ε, να χρειάζεται παρέμβαση από τους Ευρωπαίους νομοθέτες με τον ε, κανονισμό αυτό για τη ρευστότητα. Όπως είπε κάποιος βουλευτής, είναι ιδιαίτερα περίπλοκο το πεδίο και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και για την υλοποίηση αυτών των πρώτων μέτρων να αντλήσουμε από όλη την συγκεντρωμένη μας εμπειρία ως τώρα. Όμως το σίγουρο είναι ότι στο ρυθμιστικό μας πλαίσιο υπάρχουν σοβαρά κενά και υπάρχει ανάγκη κάπως να καλυφθούν. Ανάγκη κεφαλαιοποίηση στην τραπεζική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως προκύπτει και από τις συστάσεις της Βασιλείας, και την, ε, τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών είναι κάτι που έπρεπε να γίνει. Η κατεξουζότητα σε αυτή πράξη λοιπόν λαμβάνει υπόψη ε, όλες αυτές τις συστάσεις και της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής και την πραγματικότητα στις χρηματοπιστωτικές ε, αγορές, τις χρηματοοικονομικές μάλλον αγορές. Να στραφώ τώρα στον κύριο Γίγκολτ και να πω ότι αυτή η κατεξοδότηση πράξη κάπως παρέκαμψε τη συμφωνία της Βασιλείας και πέρασε από τις υπηρεσίες της Επιτροπής. Αυτό ήταν το σημείο αφετηρίας μας, ε, η μελέτη της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών. Βάσει αυτών των πορισμάτων εργαστήκαμε στις υπηρεσίες της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να πω ότι τεχνική ανάλυση που έγινε από την Ευρωπαϊκή Αρχή για τα ε, καλυμμένα ομόλογα. Αυτά είχαν υψηλή ρευστότητα σε πολλές περιπτώσεις. Και εκεί υπήρχε πολύ μεγαλύτερη ρευστότητα από κάποιες περιπτώσεις δημόσιου κρατικού χρέους. Οπότε με την πρακτική μας ανάλυση είδαμε ότι τα καλυμμένα ομόλογα έπρεπε να τύχουν καλύτερες μεταχείρισεις από ό,τι στην ανάλυση και στη μελέτη της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών. Παρόμοιο ε, το συμπέρασμα για κάποια από τα στοιχεία της τυπλοποίηση. Ξέρουμε ότι η συμφωνία της Βασιλείας και συστάσεις της ΕΜΠΑ, της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών, για τα ε, ενυπόθηκα ομόλογα και τις, ε, τους τίτλους έχουν ε, πιο ευνοϊκή μεταχείριση. Υπάρχουν όμως και άλλα προϊόντα που έχουν καλά αποτελέσματα. Οπότε με σκοπό την τιτλοποίηση και ως εναλλακτικό μέσο χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας θεωρήσαμε ότι χρειάζεται να, δοθεί διαφορετική, να τύχουν διαφορετικές μεταχείρισεις στην κατεξοδότηση πράξη κάποια μέσα τιτλοποίησης που μπορεί να επιτρέψουν να δημιουργηθεί ζήτηση για τέτοιου είδου ε, στοιχεία ενεργητικού και προκειμένου να παραμείνουμε στα πλαίσια της προληπτικής ε, ε, καθοδήγησης από τη Βασιλεία. Αυτές είναι οι δύο βασικές διαφορές για την ευνοϊκότερη μεταχείριση των καλυμμένων ομολόγων και της τυπλοποίησης. Βεβαίως να τονίσω, όπως είπατε, ότι για κάποιες συνεταιριστικές τράπεζες, τράπεζες αποταμίευσης και το τι μεταχείρισεις έτυχαν αυτές την καταξιοζότηση πράξη, νομίζω το ζωμί εδώ είναι ότι η Συμφωνία της Βασιλείας ε, σχεδιάστηκε και σταθμίστηκε για να εφαρμοστεί σε ένα μικρό αριθμό ε, πολυεθνικών τραπεζών, σε ε, ενοποιημένο μόνο επίπεδο, και για τράπεζες που τη ρευστότητά του την έχουν στις ε, χώρες, όλες τις χώρες όπου ισχύει η Συμφωνία της Βασιλείας. Άποψη λοιπόν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν ότι το να βάλουμε τόσο στενά όρια σαν ζουρλομανδία για τα ε, κάλυψη της ρευστότητας θα ήταν πάρα πολύ ε, πιεστικό θα έπρεπε να αφήσουμε κάποιο περιθώριο τυπλοποίησης για κάποιους που είχαν ήδη πολύ καλά αποτελέσματα στην Ευρώπη και να, να εφαρμοστεί αυτός ο δείκτης για όλες τις τράπεζες στην Ευρώπη με διαφορετικό τρόπο, δηλαδή να λάβουμε υπόψη την διπλή πραγματικότητα. Αυτή ήταν η συνολική μας προσέγγιση για τις προσαρμογές που έγιναν στην αναγνώριση κάποιων ιδιαίτερων χαρακτηριστικών. Να ολοκληρώσω Σα στις παρατηρήσεις του Σας διαβεβαιούμε ότι η κατεξοδότηση πράξη σε καμία περίπτωση δεν ε, υπερέχει των διατάξεων επίπεδου 1. Και αυτές ισχύουν στο βαθμό που αφορούν υποχρεώσεις του κανονισμού κεφαλαιακών απαιτήσεων ουσιαστικά μεταφράζονται η μορφή και το περιεχόμενο των υποχρεώσεων κάλυψης ρευστότητας σε ένα ευρύ φάσμα κανόνων που έχει γίνει σε διεθνές επίπεδο και που έχει συστήσει και η ΕΜΠΑ. Η κατεξουσιοδότηση πράξη λοιπόν ουσιαστικά μεταφράζει τις απαιτήσει για υποβολή εκθέσεων της, ε, του κανονισμού για τις κεφαλαϊκές απαιτήσει. Δεν αλλάζουν σε καμία περίπτωση οι υπόλοιπες υποχρεώσεις που προβλέπονται από τις ε, διατάξεις ρευστότητα του κανονισμού κεφαλαϊκών απαιτήσεων. Με την ΕΜΠΑ συνεργαζόμαστε για να έχουμε ένα ενιαίο πλαίσιο υποβολής εκθέσεων που να βασίζεται ή να αντικατοπτρίζεται τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων για τη ρευστότητα, όπως προκύπτουν από τον κανονισμό και όπως τώρα μεταφράζονται από την κατεξουσιοδότηση πράξη. Προσπαθούμε να ετοιμάσουμε τέτοια πλαίσια, πρότυπα, που ελπίζουμε να είναι έτοιμα ως τον ερχόμενο Απρίλιο, και θα δώσουμε έξι μήνες στις εποπτικές αρχές και τους υπεύθυνους φορείς για να χρησιμοποιήσουν αυτά τα πλαίσια, αυτά τα μοντέλα και να αρχίσουν να τα εφαρμόζουν στην υποβολή εκθέσεων. Γι' αυτό για την κατεξοδότηση πράξη για τον δίκτυο κάλυψη ρευστότητα προτείναμε τον Οκτώβριο του 2015 ε, θέση σε ισχύ ώστε να προλάβουν όλοι να συμμορφωθούν με αυτό το νεμεθότημα βασική δουλειά θα είναι για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τις συνεταιριστικές τράπεζες. Αλλά εφόσον χρειάζεται να σας απαντήσω ξεχωριστά για τέτοια θέματα. Σας ευχαριστώ πολύ και νομίζω ότι τώρα μπορώ να δώσω το λόγο και πάλι στον εισηγητή. Δεν έχει άλλο σχόλια. Πολύ ωραία. Μάλιστα. Όπως ξέρετε το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μέχρι τον 12 Ιανουαρίου του 2015 μπορούν να αντιδράσουν γιατί 10 είναι Σάββατο αλλά θα πρέπει να μέχρι αύριο να κάνουμε μια πρώτη ανταλλαγή απόψε έως τώρα δεν έχουν γίνει τέτοια σχόλια δεν, έχουν, δεν έχει λάβει γραμματεία τέτοια σχόλια Νομίζω λοιπόν ότι μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη να σχολιάσω μόνο κάτι που είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το οποίο εμείς στο ε, Κοινοβούλιο θεωρούμε ότι τη συμφωνία δεν αποτελεί νομοθετικό σώμα. Δικός μας ρόλος είναι να αξιολογήσουμε και να εφαρμόσουμε κατάλληλο τις συστάσεις αυτές βάσει της δημοκρατικής εντολής που έχουμε λάβει. Στο 3 υποβολή εκθέσεων αναχώρα που δεν είναι πράξη κατά εξουσιοδότηση, αλλά έκθεση που ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 30 Οκτωβρίου για τις οικονομικές συνέπειες των απαιτήσεων υποβολής εκθέσεων αναχώρα που ξεκίνησε με τα πρωτοβουλία του Κοινοβουλίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε ως καθήκον να εξετάσει και να αξιολογήσει κατά πόσον αυτές ε, οι εκθέσεις αναχώρα είχαν αρνητικές επιπτώσεις στην οποία περίπτωση θα χρειάζονταν τροποποίηση της νομοθεσίας ή κατά πόσον δεν υπάρχει αρνητικός αντίκτυπος. Από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει αρνητικός αντίκτυπος, αλλά Ας αξιολογήσουμε την έκθεση της Επιτροπής και να δώσουμε και πάλι το λόγο, α, συγγνώμη, πρώτα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μας παρουσιάσει τα πορίσματά της. Thank you. Unfortunately... Ευχαριστώ. Δυστυχώς ο τμήματάρχης προϊστάμενος μου, ο Γερμαν Χόιερ, θα αργήσει λίγο γιατί είναι απασχολημένο σε άλλη επιτροπή. Θα σας δώσω εγώ όμως μια σύντομη περίληψη των συμπερασμάτων και των πορισμάτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ό,τι αφορά την δημοσιοποίηση πληροφοριών αναχώρα με βάση το άρθρο 89 της 4ης Οδηγίας Κεφαλακών Απαιτήσεων. Το άρθρο 89 της ε, οδηγίας αυτής ε, απαιτεί από τις τράπεζες και τις επιχειρήσεις επενδύσεων να ε, δημοσιοποιούν σε αιτήσια βάση και για κάθε χώρα χωριστά κάποια στοιχεία. Δυστυχώς φαίνεται ότι δεν λειτουργούν οι διαφάνειες. Το άρθρο 89 λοιπόν απαιτεί από τα ιδρύματα να δημοσιοποιούν στοιχεία για τα κέρδη τους, τους φόρους επί των κερδών και τις επιδοτήσεις, τις δημόσιες επιδοτήσεις που λαμβάνουν. Και αυτό αναχώρα. Η έκθεσή μας ε, στηρίχθηκε στο άρθρο 89, παράγραφος 3 της Οδηγίας Κεφαλαϊκών Απαιτήσεων, ΟΚΑ, που ζητά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προβεί σε μια γενική αξιολόγηση των πιθανών αρνητικών οικονομικών αντικτύπων και συνεπειών του CBCR. Και μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2014 έπρεπε να δημοσιεύσουμε τα συμπεράσματά μας. Και μάλιστα επιταχύναμε κάπως το χρονοδιάγραμμα για να ε, εγκριθεί αυτό το ζήτημα από την προηγούμενη Επιτροπή. Στόχος της αξιολόγησης ήταν να διαπιστώσουμε κατά πόσο υπάρχουν σημαντικές αρνητικές οικονομικές συνέπειες ε, της υποχρέωσης δημοσιοποίησης πληροφοριών αναχώρα. Αν ε, εντοπίζαμε τέτοιες αρνητικές συνέπειες θα έπρεπε να τροποποιήσουμε τις υποχρεώσεις ή και να τις ε, καταργήσουμε. Το άρθρο δεν έχει τεθεί πλήρως ακόμη σε ισχύ. Ήταν ουσιαστικά μια προκαταρκτική ανάλυση και πολύ διορατική, ζητήσαμε με διαβουλεύσεις και έρευνα τις απόψεις των ενδιαφερομένων. Μάλιστα, καταρτήσαμε και μία οικονομετρική ανάλυση για να εξετάσουμε τα αποτελέσματα και της βελτίωσης ε, ε, της ε, υποχρέωσης αυτής ε, και, το, και κυρίως επιπτώσει στη διαχείριση κερδών, εσόδων και επίσης τη δυνατότητα εμπιστευτικής χορήγησης τέτοιων πληροφοριών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από τις μεγαλύτερες εταιρείε. Τα συμπεράσματα δεν διαπιστώνουν σημαντικές αρνητικές οικονομικές συνέπειες. Υπάρχουν κάποιες θετικές συνέπειες Επαναλαμβάνω, είναι μια προκαταρκτική αυτή η εργασία και έγινε εκ των προτέρων για τη διαφάνεια θετικές συνέπειες, για τη λογοδοσία του χρηματοπιστωτικού τομέα. Από τις πληροφορίες ε, και τις απόψεις των ενδιαφερομένων ε, αναμένεται από τους ε, επενδυτές να ε, λαμβάνουν πιο τεκμηριωμένες αποφάσεις, όντας καλύτερα κατατοπισμένοι και επίσης να ζητούσε μεγαλύτερη λογοδοσία και επίσης ε, ε, τα Ιδρύματα θα κάνουν καλύτερη διαχείριση των κινδύνων και θα περιοριστεί έτσι και ο κίνδυνος σκανδάλων όπως αυτά που είχαμε. Οι ενδιαφερόμενοι που είχαν θετική άποψη θεώρησαν ότι αυτή η υποχρέωση θα προσελκύσει επενδυτές και πελάτες και θα ενισχύσει τη διαφάνεια. Σε ό,τι αφορά την οικονομετρική ανάλυση, η βελτιωμένη δημοσιοποίηση, που είναι ο βασικός στόχος αυτής της υποχρέωσης δημοσιοποίησης, θα έχει θετικές συνέπειες, όπως μείωση του κόστους ε, του, του κεφαλαίου, του ίδιου κεφαλαίου, μείωση, ε, ε, μάλλον βελτίωση της διαχείρισης των εσόδων, μείωση της δυνατότητας διαχείρισης των εσόδων και καλύτερη λογοδοσία η πολέμη της πρότασης, για όσοι είχαν αμφιβολίες για τη δημοσιοποίηση αυτή, έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου προς τη δυνατότητα παρεξήγησης ως προς τα δημοσιοποιημένα στοιχεία και στην, ε, στον κίνδυνο να αυξηθεί το γραφειοκρατικό άχθος, η γραφειοκρατία. Επίσης, ε, δεν τάχθηκαν κατά της ε, διαφάνειας, αλλά ζήτησαν περισσότερες καθοδηγήσεις για το συγκεκριμένο περιεχόμενο των προς δημοσιοποίηση πληροφοριών. Σας ευχαριστώ. Τώρα να δώσουμε το λόγο στον εισηγητή. Ο κύριος Κάρας. Αν θέλει να πάρει το λόγο. Πρόεδρε, Στη μία πλευρά έχουμε τη διαφάνεια που στα φορολογικά ζητήματα ενισχύεται και απαιτείται από τους πολίτες και με το βήμα αυτό και πάλι ενισχύεται η εμπιστοσύνη στις τράπεζες. Αλλά υπάρχουν και δύο θέματα τα οποία θέλω να τα θέσω. Στην έκθεση αναφέρεται ότι διάφοροι ενδιαφερόμενοι φορείς θα ήθελαν επιπρόσθετη υποστήριξη σε ό,τι αφορά τα λεπτομερή περιεχόμενα το θεμάτων της έκθεσης. Είναι πολύ γενική αυτή η διατύπωση. Υπάρχει λοιπόν κάποια επιπρόσθετη υποστήριξη. Θα υπάρχει δυνατότητα τέτοια. Και αν ναι, πώς θα διαμορφωθεί αυτή η δυνατότητα. Δεύτερον, Πολλές τράπεζες ε, δρούν διασυνοριακά σε ευρωπαϊκό επίπεδο πλέον. Και σε κάθε χώρα πρέπει να δημοσιεύουν τα ίδια περιεχόμενα. Ωστόσο αυτό συμβαίνεται με διαφορετικά templates, με διαφορετικά πρότυπα. Και αυτό είναι αντιφατικό. Τα ενιαία τέτοια πρότυπα θα έδιναν καλύτερη συγκρισιμότητα. Γιατί έτσι κι αλλιώς υπάρχουν πολλές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών. Αυτό το επιπρόσθετο βάρος, φορτίο, έχει παρατηρηθεί. Υπάρχουν σκέψεις από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την υποστήριξη της ΕΠΑ να βρεθεί ένα ενιαίο τέτοιο πρότυπο, να υπάρχει μια απλούστευση για την καλύτερη συγκρισιμότητα και για την πρώτερη αυτή παρατήρηση για τη Βασιλεία καταρχάς. Θα ήθελα να πω το εξής. Υποστηρίζω ότι η Βασιλεία δεν είναι νομοθέτης. Αυτό που θα ήθελα να υπογραμμίσω είναι το εξή, ότι ο συντονισμό των κρατών μέλων των εκπρόσωπων της, ε, ε, των κρατών μελών γίνεται ενισχυμένα στην Επιτροπή της Βασιλείας. Με την υποστήριξη των κρατών μελών στην Επιτροπή της Βασιλείας δημιουργείται ένα πρότυπο για το Κοινοβούλιο, το οποίο εμείς καλούμαστε να το διορθώσουμε. Παρά το γεγονός ότι συμμετείχε η Ευρώπη και εδώ ο συντονιστικός ρόλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι τεράστιος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να συντονίσει τα κρατημέλη στην Επιτροπή της Βασιλείας και στη διαδικασία της Βασιλείας. Έχει υποχρέωση υποβολής αναφοράς στο Κοινοβούλιο είμαστε και εμείς μέλη της Βασιλείας, δεν είμαστε διορθωτικός ε, μηχανισμός μετά την ε, έγκριση στη Βασιλεία, Θα το διευκρινίσουμε αυτό. Ευχαριστώ. Thank Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, και γι' αυτό το λόγο η, Επιτροπή μας θα ξεκινήσει μια έκθεση ακριβώς σε ό,τι αφορά τη σχέση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα διεθνή αυτό αυτά φόρουμ και χρειάζεται δημοκρατική λογοδοσία. Είναι ένα από τα θέματα που θέσατε ο κύριος Ούντο Μπούλμαν, ο Σκιώδης. Ναι, θα ήθελα και πάλι να υποστηρίξω τον Ότμαρ για τα συμπεράσματά του, αλλά να ευχαριστήσω και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την έκταση. Και ιδιαίτερα θα ήθελα να συγχαρώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί ε, επέλεξαν την Coopers ως εξωτερικούς ε, συμβασιούχους για την εξωτερική αυτή ανάλυση. Τα πρώτα απορίσματα δίνουν την εντύπωση ότι αυτοί οι τύποι ξέρουν ακριβώς για το τι μιλάνε. Καταλαβαίνω την πολιτική διάσταση των ε, εκθέσεων αναχώρα. Τούτου λεχθέντους θα ήθελα να τονίσω το εξής. Αν μου επιτρέπετε να συνοψίσω του το γύρο τραπέζης. Και αυτοί που οι Pricewaterhouse Coopers επιβεβαιώνουν η εντύπωση ότι ενώ το ενδιαφέρον είναι περιορισμένο στην παρούσα φάση, θα αυξηθεί σταδιακά. Ναι, αυτή είναι και η δική μου εντύπωση, ότι θα είναι όλο και πιο σημαντικές αυτές οι εκθέσεις αναχώρα. Θα θεωρούνται ως ένα κανονικό μέσο και η Επιτροπή μας καλά έκανε και επέμεινε στις διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κυρίως με το Συμβούλιο που στην αρχή δεν του άρεσε καθόλου η ιδέα αυτών των εκθέσεων αναχώρα. Καλά κάναμε λοιπόν και επιμείναμε προκειμένου να υπάρχει μια νέα πραγματικά φρέσκια νομοθεσία. Μια νέα πνοή. Τέλος. Αυτό που προτείνουν οι ενδιαφερόμενοι φορείς από πλευράς του κοινού. Θα ήθελα να το ενισχύσω αυτό και να το θέσω στην ημερήσια διάταξη. Βλέπουμε ήδη ότι οι εκθέσεις αναχώρα θα έχουν ευεργετικά αποτελέσματα και αυτό θα πρέπει να διευρυνθεί για όλους τους, όλες τις ε, πολυεθνικές εταιρείες, όχι μόνο στον κλάδο αυτό. Αυτό λοιπόν είναι το δίδαγμα αυτών των εβδομάδων. Θα ήθελα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας υποβάλει μια σχετική πρόταση το συντομότερο δυνατόν. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Για τους συντηρητικούς και μεταρρυθμιστές, κανείς, Άλντε, ούτε, Γκουε, ο κύριος Για τα συμπεράσματα, τα πορίσματα αυτής της μελέτης. Νομίζω φαίνεται επανάληψη περί τι αυτό. Προφανώς έλειπε το στοιχείο της διαφάνειας στη λειτουργία των αγορών και των οίκων και ούτω καθεξής. Το πρόβλημα κατά με είναι ότι έχουμε επικεντρωθεί περιβολικά σε ένα σενάριο που είναι το ε, σενάριο της φυσιολογικής λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος, του όλου συστήματος και τελικά ε, παραβλέπουμε λίγο το πραγματικό πρόβλημα. Ακριβώς η κρίση, του επίκεντρό της δεν το είχε σε αυτό το σύστημα κανονικής λειτουργίας, αλλά σε αυτά που συνέβαιναν εκτός του φυσιολογικού συστήματος, εκτός των ισολογισμών των, των ισολογικών των τραπεζών, εκτός των στου φυσιολογικού παραδείσου και ούτω καθεξής. Εκεί λοιπόν πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μα. Γιατί Αυτές οι οικονομικές μελέτες τελικά δείχνουν κάποια συμπεράσματα κάποια αποστατικά, αλλά λίγο αυτονόητα και περιτά τελικά. Ευχαριστούμε για τους πράσινους. Ευχαριστούμε την Επιτροπή και την PricewaterhouseCoopers για αυτή την εξαιρετική ε, συμβολή στην περισσότερη δικαιοσύνη, στη φορολογική δικαιοσύνη στην Ευρώπη. Είμαι λίγο επιφυλακτικό όμω. Πώς ανατέθηκε αυτή η μελέτη στην Βαταχάουσκούπα, Η περίληψη που έχετε δημοσιεύσει δείχνει μια προσέγγιση πολύ καλά εξισορροπημένη και είναι και θετική είδηση ότι από το χρόνο στην Ευρώπη θα υπάρχουν αναχώρα δεδομένα για όλες τις τράπεζες. Αυτό είναι ένα μεγάλο βήμα πρόοδου και ήδη πολλές φορές στο Κοινοβούλιο είχαμε τη συζήτηση όπου θα πρέπει να επεκταθεί αυτή η υποχρέωση σε περισσότερους τομείς, όπως έλεγε ο Ούντο. Έχω όμω δύο ερωτήσει προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εάν αυτά τα πλεονεκτήματα που θα προκύψουν από το μεγαλύτερο βαθμό διαφάνειας για τους συμμετέχοντες στην αγορά, αλλά Όπω φαίνεται και από την αποτίμησή σα, αν αυτά ισχύουν για τι τράπεζε, τι θα γίνει με του υπόλοιπου τομεί. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα βασιστεί σε αυτή την πρόταση για να κάνει κι άλλε για του υπόλοιπου τομεί, διότι τα περισσότερα επιχειρήματα που προβάλλονται θα μπορούσαν να ισχύουν και για άλλου τομεί. Έπειτα, για τα δεδομένα που ε, για το 2014 σε βάση εμπιστευτική. Ήδη έχετε τα δεδομένα στα χέρια σας. Σκοπεύετε να ζητήσετε από τις υπεύθυνε αποστέλουσες αρχές αν συμφωνούν με τη δημοσίευση των δεδομένων. Προφανώς δεν μπορείτε να το κάνετε από μόνοι σας, αλλά μπορείτε να ζητήσετε τη κατάθεσή τους. Αυτό θα αυξήσει επίσης τη διαφάνεια. Και τέλος, Ήθελα να μου πείτε πότε θα δημοσιευτούν για πρώτη φορά δεδομένα. Πότε να περιμένουμε για πρώτη φορά να δούμε αναχώρα δεδομένα για τον τραπεζικό κλάδο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Η FTD. Ωραία. Είναι σαφές δεν προβλέπεται νομοθετική πρόταση για τι υποχρεώσει υποβολή εκθέσεων. Ε, να προχωρήσουμε. Με συγχωρείτε να δώσει μια γρήγορη απάντηση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, θα έπρεπε να περάσουμε στο επόμενο σημείο, αλλά για ένα-δύο λεπτά, αν θέλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, άντε ας πάρει το λόγο. Πολύ σύντομα ίσως να απαντήσω αντίστροφα, με την αντίστροφη σειρά. Για την τελευταία ερώτηση για το πότε θα διατεθούν τα νέα δεδομένα, νομίζω από το δεύτερο εξάμεινο του 2015. Η υποχρέωση ισχύει από 1η Ιανουαρίου 2015, οπότε το δεύτερο εξάμεινο. Ως προς το ερώτημα για το αν αυτές οι υποχρεώσεις θα επεκταθούν και σε άλλους κλάδους του δεν μπορούμε να απαντήσουμε εμείς. Είναι όμως κάτι που θα μας αποσχολήσει και το έχουμε ξανακούσει. όσο για το τι σκοπεύουμε ή μπορούμε να κάνουμε για να υπάρξει μεγαλύτερη σαφήνεια για τα στοιχεία που θα πρέπει να υποβάλλονται στις εκθέσεις, τώρα βρισκόμαστε στη φάση όπου έχουμε κάνει την καταγραφή μας και υπολογίζουμε ότι θα υπάρξουν ωφέλη, όμως τα ωφέλη αυτά αυξάνονται εφόσον υπάρχει μεγαλύτερη σαφήνεια. Γι' αυτό πρέπει τώρα να σκεφτούμε ποιο θα είναι το επόμενο βήμα. Θα χρειαστεί κάποια δράση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κάποια δράση από τον ίδιο τον κλάδο, εάν αυτή η υποχρέωση υποβολής εκθέσεων δημοσιοποίησης πληροφοριών χώρα μάλλον επεκταθεί και σε άλλους κλάδους, θα αλλάξει κάπως η ισορροπία, οπότε θα το ξαναδούμε. Ευχαριστούμε να περάσουμε στο τελευταίο αλλά όχι λιγότερο σημαντικό σημείο η εξουσιοδοτή πράξη και εκτελεστική πράξη για τι συνεισφορέ ε, στον ενίο μηχανισμό εξυγίανση βάσει τη οδηγία για την ανάκαμψη και την εξυγίανση των πιστοτικών ιδρυμάτων. Όπω ήδη έχουμε πει, ε, κάποια μέλη τη διαπραγματευτικής ομάδα ε, συμπεριλαμβανομένου ημού, εμού, του ιδίου μαζί με την Ιταλική Προεδρία συζητήσαμε στις 5 Νοεμβρίου το θέμα ακριβώς αυτό λάδουμε γνώση της εκτελεστικής πράξης για τον ενιαίο μηχανισμό εξυγένσης, όπως συζητήθηκε στις ομάδες εργασίας του Συμβουλίου, και αποφασίσαμε να παραμείνουμε σε επαφή, ώστε να συμβαδίσουν οι δράσεις των δύο θεσμικών οργάνων ως προς τα δύο αυτά θέματα. Βρίσκονται ακόμη σε πρώιμα στάδια στις συζητήσεις τους και τα δύο θεσμικά όργανα, το Συμβούλιο και η Επιτροπή δεν έχουν ζητήσει λόγου χάρη από το Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο να εκφράσουν αντίρρηση ή όχι για την κατεξοδότηση πράξη. Εγώ επιμένω αυτά τα δύο στοιχεία να εξεταστούν ως μέρος του πακέτου. Βεβαίως είναι δική μας αρμοδιότητα βάσει των όσων ισχύουν για, τα, για τις κατεξοδότηση πράξης να τοποθετηθούμε. Να ξαναπώ ότι ως Επιτροπή θεωρούμε ότι δεν έχουμε ενημερωθεί επαρκώς για τις εξελίξεις, για την εξοδέτηση πράξη τα μαθαίνουμε από τα παρασκήνια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή από τα κράτη-μέλη και πρόκειται για πάρα πολύ σημαντικές και ευαίσθητες συζητήσεις. Δεν υπάρχει όμως επίσημη ενημέρωση για την ώρα προς την Επιτροπή μας. Κάτι που ε, καλό θα ήταν να μην επαναληφθεί στο μέλλον. Να δώσω το λόγο στον Γκούναρ Χόκμαρκ, τον ε, εισηγητή. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και αυτά που μας είπατε είναι πολύ σημαντικά και μας βρίσκουν όλους σύμφωνος. Είναι σημαντικό ε, να λάβουμε υπόψη ότι οι εφαρμοστικές ε, πράξεις για τον ενιαίο μηχανισμό εξυγίασης θα πρέπει να συνδέονται με τις κατεξοδότησες πράξεις ε, του κανονισμού για την ανάκαψη και την εξυγίαση χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, γιατί είναι αλληλένδετα τα δύο θέματα. Είναι σαν δίδυμες πράξεις. Θα πρέπει λοιπόν από κοινού να εξετάζονται για πολλούς και διάφορους λόγους. Έχουμε το ενίο εγχειρίδιο κανόνων καταρχήν, οπότε οι ίδιοι κανόνες πρέπει να ισχύουν και στην Ευρωζώνη και στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι σημαντικό να λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι έχουμε ήδη 11 Νοεμβρίου. Και και λόγω της νομοθεσίας μας αλλά και λόγω της πραγματικότητας είναι σημαντικό και τα δύο νομοθετήματα να τεθούν σε ισχύ από την 1η Πρώτου 2015. Είχαμε συνεδρίαση της Επιτροπής μας τον Ιούλιο και εκεί είχα επισημάνει την ανάγκη και η κατεξουδότηση πράξης και οι εφαρμοστικές πράξεις να ευθυγραμμίζονται με τα νομοθετικά κείμενα. Δηλαδή, απαιτείται αναλογικότητα και μια προσέγγιση που θα στηρίζεται στον κίνδυνο. Και μια και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέφερε κάποιες αλλαγές, θα πρέπει να το εξετάσουμε. Πάντως είπα στις συζητήσεις ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τα αιτήματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τις απόψεις των πολιτικών ομάδων στη γενικότερη συζήτηση. Επισήμανα ότι ακόμη και μικροαλλαγές μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Και είναι κρίμα που τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως περιμέναμε. Γιατί είναι θέμα πολιτικού γοήτρου και κύρους. Και σε τελική ανάλυση και κατεξοδότηση πράξεις και εφαρμοστικές πράξεις ε, διατρέχουν τον κίνδυνο να μην τεθούν σε ίσια εγκαίρος εξαιτίας αυτού του πολιτικού θέματος. Κάτι που είναι απευκταίο. Πιστεύω ότι η εφαρμοστική πράξη θα πρέπει να συνάδει με την κατεξουσιοδότηση πράξη. Και φυσικά να έχουν και οι δύο μορφή και περιεχόμενο που να μπορούν να γίνουν δεκτά από μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και να επαναλάβω κάτι που αναφέρθηκε προηγουμένως. Είναι σημαντικό και επιτακτικό να περιορίσουμε τη σημασία ή το μέγεθος των παραγόγων. Και αυτό μπορεί να γίνει εύκολα κατά τη γνώμη μου. Και θα έχει μεγάλη σημασία και για την εφαρμοστική πράξη που αφορά τον ενιαίο μηχανισμό εξυγίασης. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να βελτιώσει κάπως επιδόσεις ό,τι αφορά το risk spread. Και πιστεύω ότι και το Συμβούλιο θα πρέπει να συνεργαστεί καλύτερα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την σταδιακή εφαρμογή και σταδιακή σύσταση του Ταμείου. Νομίζω ότι Ακριβώς επειδή πρόκειται για χαρτογραφημένα είδατα, για γνωστά πράγματα και για συζήτηση που έχουν ήδη, για συζητήσεις που έχουν γίνει ήδη γίνει, δεν είναι τόσο δύσκολο. Το είχαμε επισημάνει και στη συνάντησή μας με την Ιταλική Προεδρία. Δεν είναι η πρώτη φορά που λέμε κάτι τέτοιο. Και είναι κρίμα που ακόμη και κάποιες μικρές αλλαγές που θα έκαναν τη διαφορά και ήταν απαραίτητες, ούτε και αυτές δεν έχουν γίνει. Και εγώ ως εισηγητής ε, για την οδηγή για την ανάκαμψη και εξηγήση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων θα ήθελα να τονίσω το, τη σύνδεση του θέματος αυτού με την εφαρμοστική πράξη. Θα ήθελα πάντως το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνουν τα δέοντα ώστε να μπορέσει και η δική μας Επιτροπή ΕΚΟΝ να εγκρίνει την κατεξοδότηση, τις πράξης. Γιατί αν δεν εγκρίνουμε τη διαδικασία στο σύνολό της, ελοχεύει ο κίνδυνος να καταψηφίσουμε και την κατεξοδότηση πράξη. Ας αποφύγουμε αυτή την πολιτική αντιπαράθεση και ας αποφύγουμε αυτή την απώλεια πολιτικού κύρου τις επόμενες εβδομάδες. Ο εισηγητής για το SRM και ο σκιώδης ό,τι αφορά το SRD, η Ελίζα Φερέ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι πολλά ήδη έχουν γίνει και μέσω ε, εσάς, Πρόεδρο, και του κυρίου Χόκμαρκ. Το πρώτο σημαντικό μήνυμα το οποίο θα πρέπει να αποστείλουμε είναι η πολιτική σύνδεση που υπάρχει μεταξύ των πράξεων κατά εξουσιοδότηση και των εφαρμοστικών πράξεων, της εφαρμοστικής πράξης. Από κοινού σε ό,τι αφορά την θετική τοποθέτηση του Κοινοβουλίου για τη θέση σε ισχύ του όλου συστήματος των εισφορών των τραπεζών από 1η Ιανουαρίου 2015. Αυτό λοιπόν προαπαιτεί πολύ προσοχή και μεγάλο επίπεδο λεπτομέρειας σε ό,τι αφορά τα θέματα αυτά, σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του κειμένου, προκειμένου να μην προκύψουν τελικά από πλευράς Κοινοβουλίου μεγάλα ερωτήματα σε σχέση με το πακέτο. Σε ό,τι αφορά την άρνηση της πράξης κατά εξουσιοδότηση. Αυτό αποτελεί μια σύνοψη ουσιαστικά των όσων ήδη έχουμε ακούσει. Σε σχέση τώρα με το περιεχόμενο της ε, πράξης, της εφαρμοστικής πράξης. Όπως είπατε δεν είναι κάτι που το Κοινοβούλιο άνετα καταλαβαίνει ότι γίνονται ακόμα πολλές αλλαγές στο περιεχόμενο των συμβολών, των συνεισφορών αυτών από πλευρά του ιστορικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φυσικά περιμένουμε μια κάποια σταθεροποίηση του κειμένου. Συμβατή και με αυτά που δηλώσαμε στο νομικό κείμενο πρώτου επίπεδου και με αυτά που γνωρίζουμε από το κείμενο του BRD. Ένα άλλο σχόλιο. Φυσικά και κατανοούμε ότι οι προσαρμογές οι οποίες έγιναν από το Συμβούλιο το νομικό κείμενο του SRM σε ό,τι αφορά στην ε, προοδευτική ενιοποίηση των τμήματων προωθεί αυτή τη λογική της αναντιστοιχίας της λειτουργίας του SRM και των συνεισφορών. Αν από το επίπεδο 1, από 1η Ιανουαρίου 2016 δηλαδή, όλες οι παλιές συνεισφορές ενοποιηθούν άμεσα και κατανεμηθούν βάσει του προφίλ αξιολόγησης κινδύνου της κάθε τράπεζας μέχρι να φτάσει το ποσό των 55 δισεκατομμυρίων που είναι το ποσό που έχει υπολογιστεί σε ό,τι αφορά τις καταθέσεις. Αυτό δεν υπήρξε λοιπόν ως ε, δυνατότητα. Έχουμε μία οκταετή περίοδο με τα παλιά τμήματα και με σταδιακή προσαρμογή τους. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι αυτό αφορά τις συνεισφορές των τραπεζών σε ό,τι αφορά τον BLRD και σε ό,τι αφορά αυτά που θα πρέπει να πληρώσουν, να συνεισφέρουν στα πλαίσια του SRM και ότι θα υπήρχε αναντιστοιχία σε ό,τι αφορά τα κράτη-μέλη όπου οι καταθέσεις είναι ποσοστιαία άνω του μέσου όρου σε σχέση με τα άλλα κρατημέλη, όπου είναι διαφορετικό το ποσοστό αυτό. Υπάρχει λοιπόν αυτό το σύνθετο στοιχείο. Το γεγονός ότι το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας έχει προτείνει έναν μηχανισμό διορθωτικό πολύ λεπτομερή, πολύ πολύ σύνθετο. Κατανοούσαμε από τη συνάντηση με το Συμβούλιο ότι αυτό βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Και επί του παρόντος θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνεχιστεί ο ανεκτός διάλογος. Να μην υπονομεύσουμε τις λεπτομέρειες του SRM και των συνεισφορών. Να μην υπονομεύσουμε αυτό που αποφασίσαμε από κοινού σε ό,τι αφορά την ε, πρωτεύουσα νομοθεσία. Τελευταίο σχόλιο, επειδή όπως είπαμε και προηγουμένως πρόκειται για χαρτογραφημένα είδατα. Τελικό σχόλιο. Αν ε, πρέπει να ψηφίσουμε στο Κοινοβούλιο θα πρέπει να ψηφίσουμε μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου την ομάδα την εβδομάδα της Ολομέλειας για να έχει ολοκληρωθεί η νομοθεσία μέχρι 1 1η Ιανουαρίου. Θα πρέπει λοιπόν στην περίπτωση αυτή να ενισχύσουμε την ανταλλαγή πληροφοριών και τη γενική συμφωνία την οποία επιθυμούμε, χωρίς όμως να υπάρχει οποιαδήποτε αρνητική συνέπεια για το συμβιβασμό αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Τώρα να δώσω το λόγο στους κοιότης. Δεν έχουμε όμως πάρα πολύ χρόνο. Παρακαλώ λοιπόν να παραμένετε στο δίλεπτο ο καθένας. Για όποιον βέβαια θέλει το λόγο. Πρώτα απ' όλα για τους φιλελεύθερους. Όχι. Τόιερ για τους Ευχαριστώ, Πρόεδρε, συνάδελφοι. Καταρχάς, οι δύο εισηγητές με σαφήνεια έθεσαν τα ερωτήματα και την κριτική τους με αποχρώσεις. Να το διευκρινίσω από πλευράς της Άλντα. Είναι ακατανόητο ότι στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το θέμα του κινδύνου δεν λαμβάνεται επαρκώς υπόψη όπως είχε ζητήσει στο παρελθόν το Κοινοβούλιο στις αποφάσεις τους. Γι' αυτό λοιπόν ερωτώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί το... η περίοδος κινδύνου είναι λιγότερο ρυθμισμένη και μικρότερη. Γιατί σε σχέση με, την, ε, με τη ΣΥΠΑ, σε ό,τι αφορά τις πυλώνες. Ο κίνδυνος υποτιμάται. Λαμβάνεται υπόψη το μέγεθος της τράπεζας. Αλλά δεν ε, είναι σίγουρο ότι αυτό αρκεί, γιατί μπορεί να υπάρχουν και μικρές τράπεζες που κάνουν συναλλαγές υψηλού κινδύνου. Γιατί? Να υπάρχει αυτή η διακριτική μεταχείριση σε σχέση με τις τράπεζες που έχουν συναλλαγές που είναι μεγάλες ε, τις τράπεζες αλλά έχουν περιορισμένο κίνδυνο στους συναλλαγές τους. Γι αυτού λοιπόν, γιατί λοιπόν δεν ε, σταθμίζεται καλύτερα στη νομική αυτή πράξη ο παράγοντας του κινδύνου. Σας ευχαριστώ. Γκουα. Ο κύριος Δεμάζιο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Το όλο νόημα αυτού του εγχειρήματο για τις τράπεζες ήταν το Ταμείο Εξυγίανσης, το οποίο ε, να διοργανωθεί σε επίπεδο 1. Και η δέσμευση να προστατευθούν οι πολίτες από ενδεχόμενη πτώχευση τραπεζών. Οι συνεισφορές των τραπεζών θα πρέπει να σε επίπεδο 1 θα πρέπει να ρυθμίζονται βάσει του κινδύνου της τράπεζας. Δεν θεωρούμε ότι αυτό διασφαλίζεται. Τράπεζες με... Σε επίπεδο 2 τώρα, οι τράπεζες με μικρότερο κίνδυνο συμπεριλαμβάνονται και τα σχετικά ιδρύματα και θα έχουν τέτοιες κρατικές εγγύησεις. Και η κατάσταση είναι η εξή. Μία τράπεζα με ψηλό κίνδυνο πληρώνει τα διπλά σε σχέση με κάποια άλλη τράπεζα σε ό,τι αφορά την κατανομή κινδύνου, το risk spread. Στη Γερμανία αυτό αφορά περίπου το 20% των ταμείων, των μισθωτικών ταμείων και υπάρχει αυτός ο ειδικός ε, ειδική ρύθμιση να μπορούν τα κράτη-μέλη να διευρύνουν αυτή τη ρύθμιση σε τράπεζες 30 δισεκατομμυρίων. Αυτό σημαίνει 10% ε, ελάφρυνση. Αυτό για προβλητικό κατά κράτη-μέλη. Μπορούν λοιπόν αυτή τη ρύθμιση για τις μικρές τράπεζες να την διαβρύνουν για τράπεζες για τράπεζες ε, πάνω από 300 δισεκατομμύρια. εκατομμύρια. Δεν καλύπτονται όμως οι τράπεζες με ισολογισμό καλύτερα από 3 δισεκατομμύρια ευρώ, αλλά με δεσμεύσεις μικρότερες από 300 εκατομμύρια μείων του ιδιωτικού κεφαλαίου του, του κεφαλαίου τους. Αυτό τι σημαίνει ότι στη Γερμανία θα ήθελα να ξέρω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι σημαίνει αυτό συγκεκριμένα. Αυτό θα πρέπει να διευκρινιστεί νομικά για την αλλαγή στη διατύπωση αυτή και τι συνέπειες έχει. you. Ευχαριστούμε. Να το ξεκαθαρίσω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι δεν κατάλαβα απολύτως διότι ε, ε λέγεται πάνω από 300 για τις καταθέσεις, όχι κάτω. Οπότε μπορεί να υπάρξει κάλυψη κάτω από τα 300 εκατομμύρια. Δεν θα επαναλάβω αυτά που είπαν οι συνάδελφοι. Ο κίνδυνος δεν έχει ληφθεί αρκετά υπόψη. Οι αριθμοί που μας δείξατε και το είδαμε και από τα δεδομένα ότι χοντρικός ότι οι εισφορές πέραν των πολύ μικρών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων βασίζονται στο μέγεθος. Η σωστός, ο σωστός υπολογισμό του κινδύνου είναι κατά προσέγγιση. Αυτό αντίκειται και στη βασική ιδέα του, της πράξης του επίπεδου, για τους κανόνες του επίπεδου 1. Γι' αυτό έγιναν και διάφορες παρατηρήσεις από τους συναδέλφους, δεν θα τις επαναλάβω, απλώς να τονίσω ότι υπάρχει ιδιαίτερος πρόβλημα με τις τράπεζες που κάνουν, που λειτουργούν προσωρινά. Και τώρα θέλουμε να δημιουργήσουμε νέες τέτοιες τράπεζες μετά την κρίση που θα εξαιρούνται από τους κανόνες των κεφαλαιακών απαιτήσεων από τους κανόνες CRR κεφαλαιακών απαιτήσεων ε, Οπότε η ερώτησή μου είναι γιατί η προσαρμογή του κινδύνου είναι τόσο χαμηλή. Ε, ε, αν δείτε και εσείς τους δικούς σας αριθμούς, δεν συνάδει με το κείμενο επίπεδου 1 και θα έπρεπε να διορθωθεί. Το κείμενο επίπεδου 1 δεν μπορεί να είναι δικαιολογία δεν μπορεί να δικαιολογεί μάλλον τις ε, προτεραιότητες της κάθε χώρας, διότι στο Συμβούλιο η λογική ήταν ότι μια χώρα έχει τράπεζες που είναι πιο επικίνδυνες από άλλη, τότε ο κανονισμός δεν καθιστά σαφές αν πρέπει να πληρώσετε περισσότερα από την προοπτική μιας χώρας, ως προς το να έχει η χώρα σας, μικρότερο, η τράπεζά σας μικρότερο κίνδυνο. Η συλλογιστική αυτή ήταν ακριβώς αυτό που θέλαμε να ξεπεράσουμε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας δυστυχώς με την κατεξοσοδότηση πράξη ακολούθησε τη λογική του Συμβουλίου που εξετάζει μόνο αναχώρα το τι συμβαίνει και όχι την σωστή ρύθμιση, αλλά με συγχωρείτε αυτό δεν είναι νομοθετήν. Ευχαριστούμε κύριος Φέρμπερ, με συγχωρείτε. Σας ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομο. Θα ήθελα να εκφράσω την εκπληξή μου. Επί εδώ και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάναμε συζητήσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πάντα θέτουμε τα ίδια θέματα, τα οποία θέσαμε και μόλις. Τα οποία μόνο περιορισμένα αναφέρονται. Κοιτώντα την τελευταία εβδομάδα πριν την έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τι έγινε στις ε, διαυπηρεσιακές διαβουλεύσεις, ε, με τους διευθυντές ε, μέχρι την συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν τεράστια η κίνηση. Άρα τι συζητάμε μεταξύ μας, αν τελικά τίποτα από αυτά που συζητάμε δεν διατυπώνεται και τελευταία στιγμή τα πασαλίβουμε, κάνουμε μαγειρέματα, μαγειρέματα όπου πραγματικά αναρωτιέμαι τι καθόμαστε και κάνουμε, αν τελικά αυτό είναι ο σκοπός. Συγκεκριμένα τώρα για τα θέματα περιεχομένου, αξιολόγηση κινδύνου. Τονίζω αυτά που είπαν οι συνάδελφοι. Βαθμιαία προσεγγίσαμε το θέμα, 75%. Αυτό που προήλθε, επειδή κοιτάξαμε από το παράθυρο, επειδή από αυτού συμφώνησε το πλειονότητα, το πλειοψηφία στην Επιτροπή, αλλά δεν επιλύει το πρόβλημα. Πάλι υπάρχει κίνδυνο. Θα πρέπει να διορθωθεί. Δεύτερον, παράγοντα, συντελεστή κινδύνου. Το έχουμε πει διάφορε φορέ. Δεν μπορούμε για του μεγάλου να καλύπτουμε 88%. Αν θέλουμε να πετύχουμε το 90% θα πρέπει να κάνουμε κάποιους συντελεστές. Τι πρόβλημα είναι, ο κίνδυνος είναι το πρόβλημα ή το μέγεθος. Εγώ θεωρώ ότι ο κίνδυνος είναι το πρόβλημα και αυτό ότι τυπώνεται και στο επίπεδο 1. Τρίτον, το είπαν και οι συνάδελφοι, δεν είναι... Είναι το Μπέρντα είναι το, η μητρική και το SRM είναι η θηγατρική νομοθεσία. Στη θηγατρική μου φαίνεται ότι τα ξεχνάμε όλα και ξεκινάμε πάλι από την αρχή. Γιατί δεν μιλάμε για τον κίνδυνο και το μέγεθος, αλλά ποια χώρα πληρώνει τι. Μα δεν είναι το θέμα ποια χώρα πληρώνει τι. Το θέμα είναι ποια τράπεζα έχει πιο υψηλό κίνδυνο. Έτσι θα αποφασιστούν οι εισφορές, όχι το που είναι η έντρα της. Και τελευταίο θέμα, σε ό,τι αφορά το φορτίο που επιβαρύνει τις τράπεζες, τις τράπεζες προώθησης. Οι τράπεζες αυτές χορηγούν χρήματα πιστώσεις βάσει εθνικής νομοθεσίας. Αυτό το θέμα θα πρέπει να επιληθεί λοιπόν και να μην κάνουμε τέτοια μεγάλη λάθη. Ναι, Μάρκο, για κοίταξε λίγο τις ε, νομοθεσίες της Βεσφαλίας, να δεις. Ο Πίτερ Σίμον να πω ότι δεν έπρεπε. Είχα πει ότι δεν θα γινόταν σήμερα συζήτηση. Αλλά το θέμα δεν είναι να προκαλέσουμε εμπόδια εδώ. Ούτε να προκαλέσουμε καθυστερήσεις, να αναχώρα. Το θέμα πρώτη Ιανουαρίου να το κάνουμε λειτουργικό το σύστημα αυτό. Χρειαζόμαστε νομική ασφάλεια. Νομική ασφάλεια θα έχουμε μόνο αν οι μεμονωμένες τράπεζες είμαστε σίγουροι δεν θα μας κάνουν μήνυση γιατί δεν υπάρχει νομική ασφάλεια για τις εισφορές τους. Το κείμενο επίπεδου 1 που βασίζεται στο άρθρο 699 και μιλάει για όλα τα πιστοτικά εντρήματα όλων των κρατών μελών. Δεν μπορώ αυτό να το υπονομεύσω με ένα κείμενο επίπεδου 2 στο άρθρο 70 του κανονισμού σε ό,τι αφορά τις διαπραγματεύσεις μεταξύ κρατών μελών, σε ό,τι αφορά το χτένισμα που θα αλλάξει τα ποσά, τα οποία θα είναι πιο υψηλό από, άλλ, από όλα τα ποσά που έχουν να κάνουν με τον κίνδυνο. θα... Με αυτό που θέλετε εσείς, με τις ιδεολογίες σας, για να μπορούμε να παρεκκλίνουμε από το άρθρο του κειμένου 1, βάσει του άρθρου 69, δημιουργεί αυτές τις ε, συνθήκες. Να παρακαλέσω λοιπόν την νομική μας υπηρεσία να ελέγξει τη νομική βάση για να μην εγκρίνουμε εδώ στο Κοινοβούλιο κάτι το οποίο εκ των υστέρων θα αποτελέσει παράνομο κείμενο. Θα είναι αντίθετο με τον νόμο. Ευχαριστώ κύριε Πρέση. Ε, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ πιστεύω ότι ήταν ε, εύκολο αυτό το θέμα. Θα το επιλύαμε στο επίπεδο 1. Και ακριβώς αντιμετωπίζουμε σήμερα τις δυσκολίες γιατί δεν το λύσαμε στο επίπεδο 1 και επιπλέον ε, επήγηκε και η επίλυση του πια. Ευχαριστώ τον εισηγητή, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ιταλική Προεδρία γιατί ανασκουμπόθηκαν ε, και αναζητούν μία λύση που θα, είναι, θα γίνει δεκτή από όλου. Και υπάρχει μια ανησυχία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε ό,τι αφορά την ενημέρωση. Γιατί είναι σημαντικό δεδομένη τη κινητοποίηση όλων των φορέων να εξασφαλιστεί απρόσκοπτη ροή πληροφοριών. Ακούσαμε από την τελευταία ε, άποψη ότι όταν υπάρχει μια νομική αβεβαιότητα δημιουργείται πρόσφορο έδαφος για παρεξηγήσεις και παρανοήσεις. Ε, κάτι που θα πρέπει να αποφεύγεται σε μια τόσο κρίσιμη ε, νομοθεσία. Και επίσης θα πρέπει να κάνουμε δίκη προθέσεων ε, στο όνομα της προάσπισης του γενικού συμφέροντος ή ειδικών εθνικών συμφερόντων γιατί το είδαμε στην Επιτροπή μας, πέραν κανονικών διαδικασιών έχουμε και κάποιες κινητοποιήσεις που κατά τη γνώμη ανταποκρινόταν περισσότερο στα συμφέροντα συγκεκριμένων τραπεζών ή συγκεκριμένων κρατών μελών εις βάρος άλλων. Και έτσι ευνοούνται κάποιες τραπεζικές δομές εις βάρος άλλων. Τώρα, σε σχέση με αυτά που γράψαμε στο επίπεδο 1, και σε ό,τι αφορά την αναλογικότητα, τη ρήτρα διασφάλισης και το σεβασμό των, τρα... εφισταμένων τραπεζικών διαρθρώσεων και την αποφυγή στρέβλωση μεταξύ τους, όλα αυτά θα πρέπει να μας βοηθήσουν να βγούμε από το αδιέξοδο και να εξασφαλίσουμε μια ισορροπία μεταξύ της αξιολόγησης του κινδύνου διαφοροποίησης και του κινδύνου αυτού καθ' αυτού. Και θεωρώ ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά κυρίως της Ιταλικής Προεδρίας, βαίνουν προς τη σωστή κατεύθυνση και ευελπιστώ ότι με βάση αυτή την πρόταση θα συμφωνήσουμε το συντομότερο δυνατό. Και τελευταίος ο μιλητής, ο Αλένα Μασούρ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συνεχίζοντας αυτά που είπε ο Βερβάς Μπέρες, θα ήθελα να πω ότι αισθανόμαστε κάποια δυσφορία όλοι για το θέμα αυτό. Γιατί ε, μερικές φορές ε, αυτές οι υποχρεωτικές εισφορές ε, φαίνεται να μοιάζουν με φορολογία, με φόρους και φυσικά στο Συμβούλιο υπάρχει ο πειρασμός και μερικές φορές και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να παίζουμε την κυρία Θάτσερ, δηλαδή φέρτε τα λεφτά μου πίσω. Δεν θέλω οι δικές μου τράπεζες να πληρώσουν περισσότερο από άλλες. Και φυσικά όλα αυτά στο όνομα του Ευρωπαϊκού Κοινού Συμφέροντο. Αυτή ήταν μια παρατήρηση που επισημάνομαι και στην πρώτη συζήτηση που είχαμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν από αρκετές εβδομάδες. Και τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας είχε απαντήσει ότι το πρόβλημα αυτό θα το λύσει με την εφαρμοστική πράξη. Αλλά για την κατεξουσιοδότηση πράξη είπε ότι θα τηρήσει αντικειμενικά και αδιαμφισβήτητα κριτήρια. Και θα πρέπει τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας αποδείξει ότι και στην εφαρμοστική πράξη και στην κατεξουσιοδότηση πράξη έλαβε υπόψη άδεια φιλονίκητα, αδιάστα κριτήρια που δεν θα εξυπηρετήσουν περισσότερο συγκεκριμένες τραπεζικές δομές και συγκεκριμένες χώρες εις βάρος άλλων, ώστε να μπορούμε όλοι να εξηγήσουμε ε, στις χώρες μας το σύστημα και να το υπερασπίσουμε ως σύστημα που υπεραμείνεται του γενικού ευρωπαϊκού συμφέροντος. Ευχαριστώ. Και τώρα θα δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στον κύριο Γερσάντ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πολλοί από τους βουλευτές εξέφρασαν την έκπληξή τους να εκφράσω και εγώ τη δική μου με τη σειρά μου διότι κατά την εξουσιοδότηση πράξη έχουν συζητηθεί σε επίπεδα άνευ προηγουμένου μεταξύ Επιτροπής και των υπόλοιπων θεσμικών οργάνων. Και δικαίω, γιατί ήταν σημαντικές. Αλλά όπως νομίζω συμφωνήσαμε την τελευταία φορά που είχαμε συναντηθεί στις 2 Οκτωβρίου και στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας, ιδίως στο σκέλος της επικοινωνίας μας με το Κοινοβούλιο, το σχέδιο πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή άλλαξε πολύ βάση των όσων μα ε, επεσήμανε το Κοινοβούλιο, κυρίω ο κ. Όκμαρ και η κυρία Φερέιρα. Με την πρώτη μορφή του κειμένου που είχαμε δει από τον ε, Ιούνιο και τον Ιούλιο. Δεν μπορώ λοιπόν να δεχτώ παρατηρήσεις του τύπου ότι λέμε ποτέ δεν λαμβάνεται υπόψη, είναι εντελώ λάθος. Βεβαίως, αυτό που ακούσαμε στο Κοινοβούλιο και σε σχέση με όσα μόλις από ο κ. Λαμασούρ είναι κάπως αντιφατικά. Φυσικά όλα όσα υπόθηκαν εδώ δεν ελήφθησαν υπόψη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα και το δικαίωμα να ε, κρατήσει αυτά που θεωρεί ότι θα οδηγήσουν σε μια εξισορροπημένη ε, εύστοχη νομοθετική πράξη. Δεν θα απηχήσει όλες τις απόψεις που θα ακούσουν εδώ μέσα. Ιδίως για τη σημασία των κινδύνων. Ως προς αυτό δεν θα πρέπει να επιμείνουμε νομίζω στην ε, καταξιοδότηση πράξη. Πρέπει ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του. Η Επιτροπή λάβει τις δικές της, αυτό κάνει και το Κοινοβούλιο. Όπως είπατε και εσείς, εδώ πρόκειται για ένα πακέτο και θα πρέπει να δοθεί σημασία που της αξίζει στην τη πράξη. Κάποια στοιχεία βέβαια ήδη συζητήθηκαν στον ε, βουλευτή από την Άλντε για τις αμφιβολίες που εξέφρασε ένα από αν θυμάται ότι τα έδωσα όλα τα αριθμητικά στοιχεία είναι διαθέσιμα όλα αυτά τα έγγραφα στο κοινοβούλιο και γι' αυτό ακριβώς νομίζω ότι ό,τι κάναμε ήταν και συνεπές και μια ορθή υλοποίηση επίπεδου 1 και παρεπιπτόντος Αυτό θα απαντούσα και στον ίδιο βουλευτή του Άλντε που έκανε λοιπόν αυτή την παρατήρηση. Να στραφώ τώρα στην εκτελεστική. Στο εκτελεστικό μέτρο. Στα εκτελεστικά μέτρα μάλλον. Εάν θυμάστε στις τελευταίες συζητήσεις μας για τα εκτελεστικά μέτρα είχα πει με βάση την κατεξοδοτήση πράξη ότι η Ευρωζώνη θα ξανά αξιολογηθεί βάσει της απέτησης 1% στην κεφαλαιοποίηση. Είπαμε ότι αυτό θα πρέπει να αντικατοπτριστεί στην κατεξοδότηση πράξη βάσει του μεγέθους, του όγκου κτλ. Αλλά στο επίπεδο 1 προβλέπεται δυνατότητα για ένα μεταβατικό καθεστώς. Και επειδή προτάθηκε να υπάρξει ένα τέτοιο μεταβατικό καθεστώς, ένα τέτοιο μεταβατικό σύστημα, εγώ τότε είχα προσφερθεί να ξαναρθώ για να συζητήσουμε όποτε θέλετε να δούμε το συγκεκριμένο θέμα. Το σχέδιο της κατεξοδότησης, με συγχωρείτε όχι, τα εκτελεστικά μέτρα κρίθηκαν μαζί με την κατεξοδότηση πράξη, ώστε ακριβώς η Επιτροπή να δείξει πόσο ε, αφοσιωμένη είναι στο στόχο που είχαμε συμφωνήσει και τα εκτελεστικά μέτρα θα κρυθούν μάλλον αυτή την εβδομάδα από την Επιτροπή όπως επί της αρχής εγκρίθηκαν στις 21 Οκτωβρίου. Θα έχετε προσέξει ότι για να διαφυλάξουμε την ενιαία αγορά, την εσωτερική αγορά, όλους τους επί της ουσίας κανόνας τους έχουμε συμπεριλάβει στην καταξιοδότηση πράξη, διότι θέλουμε τραπεζική ένωση και χώρος της να έχουν ε, πολύ λίγο περιθώριο να παρακάμψουν τους κανόνες. Γι' αυτό κατά 99% οι κανόνες συμπεριλαμβάνονται στην κατεξοδότηση πράξη. Και αυτό ήλπιζε να το καλωσορίσει το Κοινοβούλιο. Το βασικό σημείο που καλύπτουν τα εκτελεστικά μέτρα είναι ακριβώς αυτή η περίπτωση παράκαμψης. Όπως σημείωσε η κυρία Φερέιρα, έχουμε φροντίσει το σύστημα να αντικατοπτρίζει το ε, βαθμό αμοιβεοποίησης των διαφορών τμήματων. Θα συμφωνεί η Επιτροπή σας ότι εάν είχε ισχύσει η αρχική μας πρόταση δηλαδή αν υπήρχε ένα ενιαίο backstop για όλα τα τμήματα, για το κάθε ταμείο δεν θα υπήρχε ανάγκη για μεταβατικό σύστημα, η αμεβιοποίηση του συστήματος θα έμενε αυτή που είναι και οι τράπεζες θα έπρεπε να τα βγάλουν πέρα μόνα τους χωρίς το μηχανισμό στήριξης. Αλλά τα πράγματα δεν είναι έτσι στην πραγματικότητα. Στα πλαίσια της νομοθετικής διαδικασίας και επειδή αυτό είναι το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων, έχουμε ένα σύστημα με τμήματα. Με μεταβατικό ε, στάδιο, με ένα βαθμό αμοιβοποίησης αυτών των τμήματων και χωρίς κοινό μηχανισμό στήριξης. Γιατί αυτό που θα αμοιβοποιηθεί από την πρώτη μέρα να είναι οι εισφορές γιατί από την οπτική γωνία των κρατών θα έπρεπε κάποια κάτι μέλη να ε, χρηματοδοτήσουν ουσιαστικά τα τμήματα κάποιων άλλων κρατομελών ενώ δεν έχουν ήδη πρόσβαση σε αυτά τα κονδύλια. Τελικά. Αυτή είναι η συλλογιστική όμως της πρότασης και κατά την άποψη της Επιτροπής υπήρχε λογική να υπάρξει κοινή ανάληψη με τις ίδιες εισφορές και το ίδιο ποσοστό με αυτό το ρυθμό ενώ αμοιβαιοποιούνται κάποια τμήματα. Αλλά όπως είπαμε, αυτή, αυτά τα εκτελεστικά μέτρα είναι του Συμβουλίου. Το Συμβούλιο θα τα τροποποιήσει όπως θεωρεί ότι πρέπει να το κάνει. Το Κοινοβούλιο έχει βεβαίως τη δυνατότητα να τοποθετηθεί χάρη στη λογική πακέτου. μπορεί λοιπόν ε, να απαντήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τεχνικές λύσεις εφόσον το ζητήσουν οι συνομοθέτες. Όμως η λογική του συστήματος που προτείνεται είναι κατά την άποψή μας ακλόνητη. και συνδέεται άμεσα με την σταδιακή αμοιβεοποίηση των τμήματων. Πρόεδρος, ευχαριστούμε μια πολύ γρήγορη απάντηση εφόσον χρειάζεται από τον εισηγητή. Γκούναρ, δεν νομίζω... ότι έχει νόημα τώρα να ξεκινήσουμε ένα εκτενή γύρω απαντήσεων. Και θα πρέπει το, κοινο... το Συμβούλιο που εξετάζει την εφαρμοστική πράξη να έχει συνεχίσει επαφές με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και ελπίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να εγκρίνουμε τα θέματα αυτά στην Επιτροπή όταν δούμε τη διαμόρφωση την οριστική της κατεξουδότησης και της εφαρμοστικής πράξης. Θα πρέπει όλες οι πλευρές να κάνουν προσπάθεια. Η Ελίζα Φερέιρα, ευχαριστώ. Απαιτείται προσπάθεια από όλους τους ενδιαφερόμενους, όπως μόλις ανέφερε ο κύριος Χακμάρκ. Και εγώ Ελπίζω ότι δεν θα γίνουν κάποιοι χειρισμοί τη τελευταία στιγμής για να έρθει σε δύσκολη θέση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Απευχόμαστε κάτι τέτοιο. Αλλά αυτό δυστυχώς θα γίνει αν δεν ε, σταθεροποιηθεί η θέση και η πρόταση για τον ενιαίο μηχανισμό εξυγίασης ε, κυρίως που φαίνεται ότι όλα ε, συνεχώς κινούνται δυναμικά. Ελπίζω πάντως να μπορέσουμε να ψηφίσουμε από εκείνο τα δύο για να παραμείνει αδιέρετο το πακέτο και να τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Πρώτη 2015. Ευχαριστώ. Ήταν πολύ κρίσιμη συζήτηση και θα ήθελα να πω στον κύριο Γκερσάντ ότι όντως ήταν ε, πρωτοφανής αυτός ο αριθμός ε, των συζητήσεων συζητήσεων και η ένταση των συζητήσεων για μια καταξιοδότηση πράξη και το εκτιμούμε ιδιαίτερως που ενέδωσε αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης χαίρομαι που πολλές απόψεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αντανακλώνται στο τροποποιημένο κείμενο. Όχι βέβαια όλες οι προτάσεις μας. Και φυσικά υπάρχουν μερικές φορές αποκλίνωσης αξιολογήσεις και εντός της Επιτροπής. Για το κατά πόσο ελήφθησαν υπόψη τα σχόλιά μας για την σωστή συνεκτίμηση του κινδύνου. Πάντως, εμείς τώρα θα πρέπει να ελέγξουμε κατά πόσο η εφαρμοστική πράξη, τώρα που θα, πάει, θα μεταβιβαστεί από την Επιτροπή στο Συμβούλιο, με την τροποποίηση μπορεί να παραμείνει στην, στην κατάσταση όπου 99% των διατάξεων εμένουν στην κατεξοδότηση πράξη διαδικασία. Γιατί υπάρχει παραλυσμός παραλληλισμός μεταξύ της κοινή ανάλυσης της αμοιβαιοποίησης και της μετάθεσης στα μοντέλα της ανάκαμψης εξηγήσεων των τραπεζών και του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού. Πάντως είναι πρόθυμη και συνεργάσιμη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το εκτιμούμε ιδιαίτερος. Το πρόβλημα μας είναι αν μας ζητηθεί για να επιταχυθεί η θέση σε ισχύ πιο νωρίς του στόχου, δεν θα δεχτούμε κάτι τέτοιο αν δεν δοθούν εχέγγυα για τη σταθεροποίηση της εφαρμοστικής, για την οριστικοποίηση, την αποκριστάλλωση της εφαρμοστικής ε, πράξης και δεν θα υπάρχει κίνδυνος περαιτέρω τροποποίησης. Από τη στιγμή που θα μας δοθεί αυτή η διαβεβαίωση από το Συμβούλιο θα φροντίσουμε και εμείς όπως είπε ο εισηγητής ε, να επισπεύσουμε τις διαδικασίες ώστε το, ζήτημα, το πακέτο να τεθεί σε ισχύ εμπρόθεσμα. Πάντως θα παρακολουθήσουμε προσεκτικά τη συζήτηση που βρίσκεται τώρα στα χέρια του Συμβουλίου και χαίρομαι για την προθυμία του Συμβουλίου να συζητήσει μαζί μας, γιατί αυτή είναι η προϋπόθεση που θέσαμε. Και πολλά από αυτά που μας είπατε είναι σωστά. Αλλά είναι και κάτι που επισήμανα εκ μέρους της Επιτροπής. Κάποια στιγμή η ροή πληροφοριών για συγκεκριμένες λύσεις που συζητήθηκαν και υλοποιήθηκαν και κάποιες ασυμμετρίες με τα δύο σχέδια. Ήταν ε, ελλειπής αυτή η ροή πληροφοριών, γιατί από εξωτερικές πηγές μάθαμε από δεύτερο χέρι κάποιες αλλαγές και κάποιες λύσεις και όχι απευθείας από την Επιτροπή το Συμβούλιο. Αυτά. Έχετε κάποιο σχόλιο για το 300? Ο κύριος, ο κύριος Δεμάζη, κύριε Γκερσάντ, έθεσε μία ερώτηση. Είπαμε ότι υπάρχει, θα δημιουργηθεί ενδεχομένω πρόβλημα στη διατύπωση του αρισμού για τα 300 εκατομμύρια. Μπορείτε να το διευκρινίσετε. Ναι, και για την τελευταία σας παρατήρηση. Κύριε Ντεμάζη, έχουμε επίγνωση του θέματος και σας διαβεβαιώ ότι αυτή η αλλαγή της τελευταίας στιγμής δεν είναι ε, η καλύτερη διατύπωση του κειμένου σίγουρα. Πάντως, ε, οι τράπεζες που έχουν κάτω από 300 σύνολο ενεργητικό, στοιχείο του ενεργητικού δεν θα υποφεληθούν από τη δυνατότητα πρόσβασης στο σύστημα. Πάντως, αν υπάρχει πρόβλημα, θα το ελέγξουν και οι νομικοί μας, γιατί μας ενδιαφέρει φυσικά η συνοχή. Θα ελέγξουν το κείμενο οι νομικοί για να αποφευθούν παρεξηγήσεις και παρανοήσεις και να δούμε αν καλύπτεται αυτή η κατάσταση. Αν δεν καλύπτεται θα δούμε ποιο είναι το εύρος του προβλήματος. Εδώ μιλούμε για έξι ουσιαστικά ιδρύματα από 400. Βέβαια όλες, όλα αυτά τα ιδρύματα βρίσκονται σε ένα κράτος μέρος το οποίο γνωρίζετε όλοι καλά. Οπότε θα το κάνουμε αυτό, θα το διευκρινίσουμε με την ερμηνεία του κειμένου. Αν δεν ευδοκιμήσει αυτή η προσπάθεια, θα ζητήσουμε από το Συμβούλιο να το διευκρινίσει στην εφαρμοστική πράξη του Συμβουλίου. Γιατί επαναλαμβάνω το πρόβλημα να κύπτει σε ένα κράτο μέλο μόνο που είναι και μέλος της Τραπεζικής Ένωση. Νομίζω ότι αυτός θα ήταν και πιο κομψό τρόπος για να επιληθεί οποιοδήποτε πρόβλημα στο Συμβούλιο δηλαδή. Ευχαριστούμε. Τώρα νομίζω μπορούμε να κλείσουμε αυτό το θέμα. Ήταν μια πολύ καλή ιδέα να προβλέψουμε αυτήν την χρονοθυρίδα, αυτό τέλο πάντων το χρόνο συζήτηση για το θέμα των ε, κατεξουσιοδότηση και εκτελεστικών πράξεων. Και τώρα περνάμε στο σημείο 4 της ημερήσιας διάταξης, ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο, Στόμα, με τον κύριο Τόμας Βίζερ. Τον βλέπω, να τον χαιρετήσω. Okay, Ας ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως. Αυτή είναι η τελευταία ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο Βίζερ. Στα πλαίσια των νομοδιοτήτων του μεταξύ άλλων, ως Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλευτικού Φορέα για την Δικυβέρνηση στον τομέα της στατιστικής, δηλαδή του ΕΣΓΑΜΠ θα μας παρουσιάσει την έκτη ετήσια έκθεση για τον ε, κώδικα ε, πρακτικής της Eurostat για τα στατιστικά δεδομένα και για το Ευρωπαϊκό Στατιστικό Σύστημα και θα σταθεί στις 11 συστάσεις της έκθεσης με προτάσεις για τις προσλήψεις και τις απολύσεις του ε, ανώτερου κλιμακίων management της Eurostat. Έτσι και αλλιώ. έχει μπλοκαριστεί τρομερή διάλογο για, τα στατιστικά θέματα. Ξέρετε ότι ακριβώ κολλήσαμε σε αυτό το σημείο και θα προσπαθήσουμε να το λύσουμε. Να δώσω το λόγο στον κύριο Βίζερ για 10 λεπτά. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Σα ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και προφανώ για το ενδιαφέρον σα ε, για την έκθεση τη ε, ΕΣΓΑ. Όπω είπατε, είναι η τελευταία φορά που έχω τη δυνατότητα να σας μιλήσω και κοιτώντας το, λόγο, το ρόλο της ΕΣΚΑΠ υπάρχει ένας μόνος σύμμαχος ε, για την ΕΣΚΑΠ στην Ευρώπη ολόκληρη, είσαστε εσείς. Υπάρχει ασφαλώς μια τάση όταν δίνει κανείς ε, σύμβουλες ε, για θέματα που αφορούν την κυβέρνηση, συνήθως υπάρχει διαφοροποιημένη άποψη, δεν το θέσω έτσι. Η αιτήσια έκθεση φετινή αφορά μόνο τη Eurostat. Ε, κάναμε την έκθεση ομοτήμων ε, της Eurostat στα πλαίσια μιας γενικότερης έκθεσης ομοτήμων όλων των εθνικών στατιστικών υπηρεσιών. Δεύτερη φορά που γίνεται τέτοια έκθεση από ομοτήμους. Όπως και στο εθνικό επίπεδο προσπαθούμε να είμαστε αρκετά συμβατή με τις εθνικές διαδικασίες. Η έκθεση λοιπόν βασίζεται στις απαντήσεις που έχει δώσει η Eurostat μετά από ένα ερωτηματολόγιο που απάντησε και κάναμε και συνεντεύξεις εκτεταμένες με τον Επιτρόπο Σέμετα και με τον Γενικό Γραμματέα της Επιτροπής. Πρώτα! και βασικό και καθησυχαστικό πόρισμα είναι ότι η Eurostat είναι μια εύρυθμα λειτουργούσα στατιστική υπηρεσία. Υπάρχουν τριβές ε, στο στατιστικό ευρωπαϊκό σύστημα, τις οποίες και αναλύσαμε εν μέρη μετά το διτό και τριπλό ρόλο της Eurostat. Είναι ένα τμήμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του δικαιώματος πρωτοβουλίας και αφετέρου να διευκρινίσουμε ότι μπορεί να θεωρηθεί εντός του ειδικού συστήματος πρίμους εντερπάρες θα έλεγαν κατά πάσα πιθανότητα. Εδώ λοιπόν ο ρόλος τους είναι πολύ πιο συναδελφικός, συμβουλευτικός σε σχέση με τις άλλες γενικές διευθύνσεις της Επιτροπής. Είναι λοιπόν αυτός ο διτός ρόλος, κάτι το οποίο ενδεχομένω να μην καταλαβαίνουν ε, επαρκώς οι εθνικές στατιστικές υπηρεσίες. Ενδεχομένω λοιπόν να πρέπει να το διορθώσουμε αυτό. Όπως και να έχει. Υπάρχει μια δυσκολία σε ό,τι αφορά τα στατιστικά στοιχεία που υπάγονται στο Ευρωπαϊκό Σύστημα των Κεντρικών Τραπεζών και που διαδραματίζουν ξεχωριστό ρόλο και σε πολλές περιπτώσεις έχουν ε, δική τους εξέλιξη. Αυτό λοιπόν το οποίο βρήκαμε είναι ότι η Eurostat εξετάζεται πάρα πολύ από τα νομικά μέσα που διατίθενται. Ενισχύθηκαν βάσει του πνεύματος του κώδικα δεντολογίας είναι εξαιρετική η δέσμευση της Eurostat σε ό,τι αφορά την ποιότητα και η χρήση της μεθοδολογίας και του κατάλληλου προσωπικού είναι επίσης ένα δυνατό σημείο. 60 συστάσεις, ή 16 συστάσεις μάλλον ε, ε, δημοσίευσαμε. Τέσσερις συστάσεις για την νομοθεσία, για την πρόσληψη και απόλυση υψηλών αξιωματούχων στη επίσης μια σύσταση νομικού, νομικής φύσεως για την ισορροπία μεταξύ της εφαρμογής της νομοθεσίας πλαισίου και των εφαρμοστικών πράξεων. Επίσης ε, έχουμε κάποιες συστάσεις για την ποιότητα, τη μεθοδολογία, τις διαδικασίες, για την διάδοση πληροφοριών, το οποίο αφορά ουσιαστικά το ημερολόγιο διάδοσης και δημοσίευσης, επίσης κάποιες συστάσεις για θέματα συντονισμού. Η Eurostat προφανώς, όπως ήθιστε στις διαδικασίες αυτές, ε, έλαβε την δυνατότητα να απαντήσει στα σχόλιά μας. Σε ένα σημείο υπάρχει διαφορετική τοποθέτηση σε ό,τι αφορά την αξιολόγησή μας και δεν μας προκαλεί έκπληξη αυτό, γιατί αφορά τις συστάσεις για την πρόσληψη και απόλυση προσωπικού. Αυτό ήταν αρνητικό. Να πω δύο λόγια για τις πρόσφατες εξελίξεις. Και πέρα από το έργο μας για την, εργασία μας για την έκθεση, ασχοληθήκαμε με θέματα με θέματα των εθνικών συστημάτων, με κάποιων εθνικών στατιστικών υπηρεσιών και με το Ευρωπαϊκό Στατιστικό Σύστημα. Πρόσφατα, το φθινόπωρο φέτος, ε, κάναμε δύο συστάσεις. Δημοσιεύσαμε δύο συστάσεις. Η μία σύσταση αφορά τη σημασία της ανεξαρτησίας της Eurostat και τη διάκρισης μεταξύ Eurostat και του Ευρωπαϊκού Συστήματος όπου υπάρχουν κάποια προβλήματα σαφής, σαφούς ε, διάκρισης των δύο συστημάτων. Ένα δεύτερο θέμα αφορούσε μια σύσταση που δημοσιεύτηκε προς τις γερμανικές αρχές για τη συμμόρφωση των ε, προσλήψεων υψηλών αξιωματούχων και ό,τι αφορά τον κώδικα τεντολογίας. Γιατί το κάναμε αυτό, γιατί στο παρελθόν ήμασταν συνήγορος ε, ισχυρών εθνικών στατιστικών υπηρεσιών και ήμασταν ε, υπέρμαχος της ανεξαρτησίας τους. Ένα θέμα, πιστεύω, είναι υποτιμημένο από πολιτικής ε, σκοπιάς. Από τη στιγμή που τα στατιστικά στοιχεία είναι ένα σταθερό σημείο στο νομικό μέσο, για παράδειγμα στο σύμφωνο σταθερότητας, σταματάνε να είναι στατιστικά στοιχεία και γίνονται πολιτικά θέματα. Πώς μπορούμε όλα να προστατεύσουμε αυτή την οικονομική διαδικασία λήψης αποφάσεων και ορισμού πολιτικών, αν η πίεση, η πολιτική πίεση στους υπεύθυνου ε, των στατιστικών υπηρεσιών είναι πολύ μεγάλη, τα στατιστικά αυτά στοιχεία δεν θα είναι εξίσου ανεξάρτητα με το επιθυμητό επίπεδο. Θα πρέπει λοιπόν τα επόμενα χρόνια να φροντίσουμε να προστατεύσουμε τον κλάδο αυτό και σε κάποιες ε, περιπτώσεις να τον ενισχύσουμε σημαντικά. Η ΕΣΚΑΠ δεν ε, δημιουργήθηκε ως αντίδραση στην στατιστική κρίση πριν από 6-7 χρόνια. Υπήρξαν σημαντικές βελτιώσεις σε διάφορα κράτη-μέλη, αλλά αν θέλετε είναι πολύ ευαίσθητη αυτή η ισορροπία. Όπως είπα και αυτή εξ αρχής, θεωρώ ότι υπάρχει μόνο ένα θεσμικό όργανο πραγματικά που είναι πραγματικός ουσιαστικός σύμμαχος της ΕΣΚΑΠ και της Eurostat και αυτό είναι το κοινοβούλιο αυτό. Να κλείσω όχι μόνο την αρχική μου παρουσίαση αλλά και την τρίτη μου θητεία στους κόλπους της ΕΣΚΑΠ. Στα τρία λοιπόν αυτά έτη ήμασταν η ανεξάρτητη φωνή προς υποστήριξη του κώδικα Δεντολογίας. Είμαι ευγνώμων για την υποστήριξη που λάβαμε τα χρόνια αυτά από το Κοινοβούλιο. Δημιουργείται και συστήνεται στην παρούσα φάση το νέο σώμα της ΕΣΚΑΠ. Ο Μάρτι Χιτιμέκη προτάθηκε ως νέο πρόεδρος από τη Φιλανδία. Είναι, είναι υφυπουργός ε, Οικονομικών στο Ελσίνκι. Μακρά και διακεκριμένη είναι η καριέρα του στην ευρωπαϊκή οικονομική πολιτική σε θέματα συντονισμού και σε πολλά άλλα ζητήματα και έχει διατελέσει ε, πολλά χρόνια πρόεδρος της Αστικής Επιτροπής του EFC. Τα μέλη που προτάθηκαν από το Συμβούλιο αναμένεται να είναι ο κ. Κόπς, Μάρτιν Γκούσμαν για δεύτερη θητεία, ο κύριος Τζοβανίνη για πρώτη θητεία και ασφαλώς θα υπάρχει προσδοκία το Κοινοβούλιο να προσθέσει εξίσου ικανά μέλη. Θα αλλάξει λοιπόν η σύνθεση τον Ιανουάριο, θα γίνει μια συζήτηση προσανατολισμού και είμαι βέβαιο ότι η συνεργασία μεταξύ τη Επιτροπή σα και τη ΕΣΚΑΠ τα επόμενα χρόνια θα είναι εξίσου θετική, ευεργετική και θερμή όπως το παρελθόν για την ποιότητα των στατιστικών δεδομένων αλλά και τη χάραξη πολιτική. Αυτή είναι η δική μου εμπειρία. Σα ευχαριστώ πολύ. σα ευχαριστώ, λέει Ευχαριστούμε για τη συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Κοινοβούλιο ήταν ανέκαθεν ε, υπέρ του ΕΣΓΑΠ, του Ευρωπαϊκού Συμβουλευτικού Φορέα, για να ενισχύσουμε την ανεξαρτησία του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος. Και φυσικά θα συμβάλλουμε και εμείς για να ολοκληρωθεί η διαδικασία στελέχωσης του ΕΣΓΑΠ, του Ευρωπαϊκού Αυτού Συμβουλευτικού Φορέα για τη διακυβέρνηση στον τομέα της στατιστικής. Δώσω τώρα το λόγο στον πρώτο μας ε, ομιλητή από το ΕΛΚ, η οποία είναι ομιλήτρια, η κυρία Γκαλπέλτς. Ευχαριστώ. Δεν θα μιλήσω ουγγρικά, γιατί με ενημέρωσαν ότι εξαιτία τεχνικού προβλήματος δεν μπορώ να μιλήσω ε, ουγγρικά παρά μόνο να ακούω ουγγρικά. Ή μπορώ. Α, μπορώ. Μάλιστα θα μιλήσω λοιπόν. Μάλλον το αντίθετο. Μπορώ να μιλήσω αλλά δεν μπορώ να ακούσω ουγγρικά. Οπότε θα μιλήσω ουγγρικά. Θα ήθελα να πω ότι οι στατιστικές πληροφορίες έχουν θεμελιώδη ρόλο στη δημοκρατική διαδικασία και στην χρηστή διακυβέρνηση. Η εμπιστοσύνη του κοινού στις ευρωπαϊκές στατιστικές ελευθερίες, το ευρωπαϊκό στατιστικό σύστημα επίσης έχει κέρια σημασία, γι' αυτό και θα πρέπει να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη του κοινού στο Ευρωπαϊκό Στατιστικό Σύστημα. Γι' αυτό και οι προτάσεις του κυρίου Βίζερ είναι πολύ θετικές γιατί μας δίνουν ένα νέο πλαίσιο λογοδοσίας. Οι στατιστικές πληροφορίες είναι καλές εφόσον είναι εύχριστες. Γι' αυτό και θα πρέπει να είναι ενημερωμένες, επικαιροποιημένες, προσβάσιμες και να στηρίζονται σε καλή παροχή πληροφοριών. Ταυτόχρονα χρειαζόμαστε αξιόπιστες, έγκυρες στατιστικές πληροφορίες, ελέγξιμες, για να στηρίζονται πραγματικά σε έγκυρα στοιχεία. Γι' αυτό και συμφωνούμε με την πρόταση ότι δεν θα πρέπει να επεμβαίνουμε στο έργο των εθνικών στατιστικών γραφείων εκτός και αν κάτι τέτοιο είναι απολύτως δικαιολογημένο. Και θα πρέπει να τους δώσουμε τα εφόδια και τεχνογνωσία ώστε να έχουμε πραγματικά στατιστικές πληροφορίες που θα είναι συγκρίσιμες, έγκυρες και χρήσιμες. Αν το ένα εθνικό στατιστικό γραφείο παρέχει παραπλανητικές πληροφορίες θα πρέπει όμως και τότε να είμαστε σε θέση να αναλάβουμε δράση για να αποκαταστήσουμε την ποιότητα της πληροφορίας που παρέχουν τα εθνικά στατιστικά γραφεία σε περίπτωση που διαπιστώσουμε παραβίαση. Θα πρέπει φυσικά να εξασφαλίσουμε την ανεξαρτησία των στατιστικών γραφείων. Γι' αυτό και ο διορισμός των επικεφαλής αυτών των γραφείων, των διευθυντών των γραφείων θα πρέπει να είναι διαφανής οι δεμοί θα πρέπει να μπορούμε να επεμβαίνουμε για να επαναφέρουμε τη διαδικασία στο σωστό δρόμο, εφόσον έχουν ε, παρατηρηθεί παρατυπίες. Θα πρέπει να ελέγξουμε το σύστημα στο σύνολό του, γιατί οι στατιστικές, τοπικές, περιφερειακές, εθνικές ή ευρωπαϊκές, θα πρέπει να στηρίζονται σε ακριβή έγκυρα αξιόπιστα, αμερόληπτα δεδομένα και ανεξάρτητα πολιτικής επιρροής. Θα ήθελα τέλος να επισημάνω ότι ζούμε σε ένα ραγδαία μεταβαλλόμενο κόσμο, γι' αυτό και χρειαζόμαστε στατιστικά συστήματα που θα μπορούν και αυτά να είναι ευπροσάρμοστα, να εγκληματίζονται στις ραγδαίες αυτές αλλαγές. Έχουμε νέους κανονισμούς, νέες νομοθετικές διατάξεις και νέες στατιστικές μεθοδολογίες που παρακολουθούν τις ταχείες εξέλιξεις. Θα πρέπει να ενισχύσουμε τον πυλώνα της αγοράς, για παράδειγμα, και να δίνουμε κάποια συνέχεια στις εξελίξεις της εσωτερικής αγοράς. Επαναλαμβάνω, θα πρέπει να είναι χρήσιμα προσιτά τα στατιστικά στοιχεία και έγκυρα πάνω απ' όλα αξιόπιστα. Επίσης, επιγραμμικές βάσεις δεδομένων είναι σημαντικές. Και ίσως σε αυτές τις βάσεις δεν θα πρέπει να έχουμε μόνο κάποια γυμνά νούμερα, αλλά και κάποιους πίνακες ή γραφικές παραστάσεις. Πάντως, σημεία αφετηρίας είναι ότι έχουμε 500 εκατομμύρια Ευρωπαίους πολίτες και ελάχιστοι από αυτούς είναι πανεπιστημιακοί. Θα μπορούν λοιπόν και αυτοί οι απλοί πολίτες να μπορούν να χρησιμοποιούν τα στοιχεία αυτά. Γι' αυτό και χρειάζονται γραφικές παραστάσεις. Ευχαριστούμε και τώρα για τους σοσιαλιστές και δημοκράτες. Σκιώδες. Εξηγητής ο κύριος Μπαγέ Ευχαριστώ Πρόεδρε, κύριε Βίζερ, το είπατε, είναι κεφαλαιόδου σημασία οι στατιστικέ ω προ την, πληροφο... την ποιότητα των πληροφοριών και την διαφάνεια που μα εξασφαλίζουν. Η διαφάνεια, η ποιότητα αυτή θα εξασφαλιστούν με την αναξαρτησία τη Eurostat. Γι' αυτό στην ανάγνωση της μελέτης σας πρόσεξα τις συστάσεις που κάνατε σε σχέση με τις προσλήψεις. Για το Γενικό Διευθυντή της Eurostat λέγεται ότι η θέση του θα πρέπει να ε, διευκρινίζεται ως προς τους όρους της ε, από την ε, νομοθεσία και να υπάρχει ανοιχτή υποβολή υποψηφιωτήτων σε σχέση με όσα διάβασα στην έκθεσή σα. Ήθελα να πάω λίγο πιο μακριά και να μου πείτε λίγο περισσότερε λεπτομέρειε για κάτι που αποσχόλησε και εμένα. Διότι και εγώ θα συμφωνήσω ότι το ε, Κοινοβούλιο μάλλον θα πρέπει να παίξει ρόλο στην ε, διασφάλιση τη ανεξαρτησία και του Eurostat και του διευθυντή τη. Και για τι δεσμεύσει που αναλαμβάνουν ε, και για τι περιπτώσει απολύσεων που δεν θα πρέπει να συμβαίνουν για λόγου πολιτικού. Ε, η τροποποίηση της διαδικασίας διορισμού λοιπόν ε, του Διευθυντή, κατά την άποψή σας πώς θα πρέπει να τροποποιηθεί. Τι μηχανισμοί πρέπει να προβλεφθούν για να βεβαιωθούμε ότι υπάρχει ανεξαρτησία του Διευθυντή και των συνεργατών του. Επίσης, στην εισήγησή σας μιλήσατε για περιορισμούς και πιέσεις ε, στους στατιστικολόγους. Ε, κατά την άποψή σας, τι πρέπει να, προβλέψουμε από την πλευρά της Επιτροπής μας για να αποφευθεί αυτό. Έπειτα, τελευταία μελέτη της Eurostat για την εξέλιξη της ένδυας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2013 που είναι ιδιαίτερα ανησυχητική. Οι αριθμοί της Eurostat δείχνουν ότι οι πολιτικές λιτότητες που εφαρμόζονται σε πολλά κράτη-μέλη, πιέζοντας τους πλέον αδυνάμους από εμά, έχουν φέρει χειρότερα αποτελέσματα. Αυτό δείχνει λοιπόν τι συμβαίνει σε σχέση με την φτώχεια και θα πρέπει όλα αυτά να τα δούμε σε σχέση και με την ε, πραγματικότητα και την καυτή επικαιρότητα και το, το, τις διαρροές για το Λουξεμβούργο, το Λουξεμβουργλίξ όπως ονομάστηκε. Οπότε θα πρέπει πιστεύετε να ε, αξιολογείτε το κεφάλαιο χώρα ένα επιχείρηση με ένα προτιμησιακό σύστημα ή να υπάρξει κάποια φορολογική εναρμόνιση ώστε να αποφύγουμε τις ε, προσπάθειες φοροδιαφυγής μια φοροδιαφύγη τελικά που ισχύει και εμφανίζεται σε όλες τις χώρες. Η Eurostat έχει στοιχεία για τα θέματα αυτά και έχει τη δυνατότητα να κάνει αυτού του είδου την ανάλυση. Ε, υπάρχουν τέτοια δεδομένα απλώ δεν δημοσιοποιούνται, δημοσιοποιούνται. Θα ήθελα λοιπόν λίγε περισσότερε διευκρινήσει. Και μια άλλη ερώτηση, λίγο τεχνικότερη, για τι ε, βασικέ προδιαγραφέ του 2000. 10 που αρχίζουν να εφαρμόζονται από το 2013 για τις επενδύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση νομίζω ότι μπορεί να πλήξουν τις κρατικές επενδύσεις και την ανάπτυξη, την οικονομική ανάπτυξη δηλαδή και την απασχόληση. Δεν νομίζω ότι η χρέωση από τις επενδύσεις των ε, αρχών τοπικής αυτοδίκησης, περιφερειακών, τοπικών ή εθνικών θα πρέπει να λαμβάνονται έτσι υπόψη. Διότι βλέπω στην εφαρμογή αυτών των προδιαγραφών δύο τεχνικά προβλήματα. Πρώτα απ' όλα πώς οι δημόσιες αρχές μέσα σε ένα έτος να αποσβέσουν μια δημόσια επένδυση. Είναι σαν να τους ε, ζητήσουμε να πληρώσουν μετρητή, μετρητής. Και ούτως ή άλλως θα είναι εξορισμού χρέος αυτό η αλλως θα ειναι εξορισμου χρέο. ενώ δεν είναι έτσι και τα δάνεια που σχετίζονται με αυτέ τι επενδύσει, ε, καταγράφονται λογιστικά ε, ως μεικτά. Ε, όμως δεν υπάρχει ε, αντιστάθμισμα στο ενεργητικό ε, με ακίνητα, με την ακίνητη περιουσία. Αυτό ε, πώς να γίνει, γιατί φαίνεται σαν να πετιέται το χρήμα και τα δημόσια κονδύλια από το παράθυρα, ενώ δεν είναι έτσι εάν δεν βρεθεί κάποιο αντιστάθμισμα. Υπάρχουμε λοιπόν σοβαρό πρόβλημα με τη μαθητολογία και τα κριτήρια που μπορεί να πλήξουν τι αρχέ τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν λέω βέβαια ότι οποιαδήποτε αρχή δημόσια θα μπορούσε να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε επένδυση χωρί καμία προφύλαξη. Όμω ο τρόπο που τα καταγράφει αυτά η Eurostat για τι δημοτικέ αρχέ περιορίζει πάρα πολύ την ελευθερία των ε, δημόσιων αρχών ως προς την ε, επενδυτική του δραστηριότητα και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Ήθελα λοιπόν και την δική σας συμβουλευτική παρέμβαση σε αυτό το θέμα. Δεν θα έπρεπε να το διαχωρίσουμε αυτό από τις ιδιωτικέ εταιρείε ε, και να λάβουμε όπως το λογιστικό αντίκτυπο που μπορεί να υπάρχει μέσα από τέτοιου είδους Και κύριε Βίζερ, Εμένα η παρέμβασή μου αυτή είναι η πρώτη σε σχέση με το δικό σας έργο, παρόλο που εσείς έχετε έρθει πολλές φορές εδώ πέρα. Οπότε ήθελα να μου πείτε στην τελευταία τριετία, είναι πολλές οι συστάσεις σας, αλλά πόσες από αυτές υλοποιήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πόσες είχαν πραγματικό και χειροπιαστό αντίκτυπο. Ευχαριστώ. Επόμενος για τους συντηρητικούς και μεταρρυθμιστές, ο κύριος Όλτσοκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, στον ε, κανονισμό για τα ευρωπαϊκά στατιστικά στοιχεία και τα ανεξάρτητα στατιστικά γραφεία σε εθνικό επίπεδο υπάρχει ένα κέριο θέμα. Μία σύντομη ερώτηση. Θεωρείτε ότι οι προδεινόμενες βελτιώσεις και τροποποιήσεις για τα απαραίτητα ε, στοιχεία διαχείρισης ε, των στατιστικών που θα εξασφαλίζουν την επικαιρότητα και την συγκρισιμότητα και τη αφήνεια θα πρέπει να δίνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ε, χάρη στις τροπολογίες αυτές θα εξασφαλίζεται η ανεξαρτησία των εθνικών στατιστικών γραφείων στην ανάληψη αποφάσεων που, που αφορούν τις διαδικασίες, τις μεθόδου στατιστικής, ε, τις προδιαγραφές και τις διαδικασίες, καθώς και την την μεταβίβαση των στοιχείων στο, Ευρωπαϊκό Γραφείο, στη Eurostat, για τις ε, ευρωπαϊκές στατιστικές πληροφορίες. Ευχαριστώ. Ο κύριος Νίλς Τόρβαλτς για την ALDE. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να πω ότι είμαστε γνωστοί για την παρέμβασή μας τις στατιστικές υπηρεσίες η πολιτική έτσι λέγεται και από στοιχεία από διάφορες ε, χώρες βλέπουμε ότι χρησιμοποιούνται για πολιτικούς σκοπούς ε, τα στατιστικά στοιχεία. Η χαρακτηριστικότερη περίπτωση είναι η Ελλάδα όπου η παραποίηση αριθμητικών στοιχείων και ο εκτελεστικός διευθυντής ε, Ανδρέας Γεωργίου αντιμετωπίζει κατηγορίες για την υπονόμευση του εθνικού συμφέροντος. Πόσο σοβαρά είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα διάφορα κράτη-μέλη ως προς αυτό, Α, κύριε Βίζερ. Ευχαριστούμε για την ΚΟΕ, ο κύριος Βιέγκας. δεν θα χρειαστεί να επαναλάβω πόσο σημαντική είναι η Eurostat για το ευρωπαϊκό οικοδόμημα συνολικά και με αυτόν τον τεράστιο όγκο στατιστικών δεδομένων για τι κοινωνικέ, οικονομικέ και πολιτικέ μα αποφάσει. Η σημασία που παίρνει η Eurostat είναι αυξανόμενη, ιδίω λόγω των αναγκών ε, που έχουν οι πολίτε και για την πρόσβαση στα βάση, στη βάση δεδομένων μέσω του διαδικτύου. Η σημασία αυτή αυξάνεται και με τη λειτουργία των θεσμικών οργάνων στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Είναι λοιπόν σημαντικό να θυμόμαστε ότι πρόκειται για μια ε, αρμοδιότητα, ένα καθήκον πολύ περίπλοκο που έχει αναλάβει η Eurostat και πρέπει να χρησιμοποιήσει συγκεκριμένη μεθοδολογία, χρονοδιάγραμμα και κριτήρια. Είναι πολύ δύσκολο να υπάρξει μια ε, πλήρης ουδετερότητα διότι τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται πάντοτε έχουν και μια πολιτική απόχρωση. Πράγμα που επηρεάζει την ουδετερότητα και την αντικειμενικότητα. Βεβαίω τα κριτήρια είναι περίπλοκα και διαρκώ υπάρχουν μεταβολέ, όπω ο νέο υπολογισμό το ΕΠ. Ε, η συζήτηση που έχουμε σήμερα σε σχέση με τα ενεργητικά. Θα υπάρξουν επιπτώσει και στου αθλητικού δείκτε που θα πρέπει να προσαρμοστούν και αυτό θα έχει επιπτώσεις και στα πρότυπα νομισματικής πολιτικής που θα εφαρμοστούν στη συνέχεια. Λόγου χάρη ο δείκτης ακίνητης περιουσίας ε, είναι ένας δείκτης τεράστιας ε, περιπλοκότητας και φοβερά ετερογενής ε, μεταξύ των κρατών μελών. Αυτός ο περίπλοκος λοιπόν χαρακτήρας που είναι έμφυτος στην ε, ε, επεξεργασία των στατιστικών δεδομένων πρέπει να γίνει αντικείμενο παρόλα αυτά εμπιστοσύνης, μια σχέση εμπιστοσύνης από την πλευρά των πολιτών. Το θέμα λοιπόν της ανεξαρτησίας της Eurostat είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το ερώτημα που θέλω να θέσω, γι, γι' αυτό μιλάει η έκθεση, είναι εάν αυτή η ανεξαρτησία έχει διακυβευτεί από τα ε, εθνικά, στα εθνικά συστήματα ή στις εθνικές υπηρεσίες ή στην Eurostat και ήθελα να μου πείτε ποιοι είναι οι συγκεκριμένοι δείκτες που μπορεί να οδήγησαν σε αυτή τη μνήμα στην έκθεση. Θα ήθελα να επικεντρωθώ επίσης και στις δημοσιονομικές περικοπές ενώ τις περικοπές των δαπανών είναι αναντήρητο γεγονός ότι η Eurostat και το Ευρωπαϊκό Στατιστικό Σύστημα μόνο να διωγκωθεί μπορεί, διότι οι αρμοδιότητες του μόνο να ενταθούν μπορούν. Πώς μπορεί λοιπόν όλα αυτά να συνάδουν με τις περικοπές που έχουν ανακοινωθεί και τι μέτρα θα πρέπει να λάβουμε στην Επιτροπή μας για να βεβαιωθούμε ότι το σύστημα συνεχίζει να λειτουργεί όπως πρέπει. Ευχαριστούμε ο κύριος Γκίγκολντ, πράσινο. κύριε Βίζερ, μία... Ερώτηση αρχικά. Θα μπορούσατε να μας βοηθήσετε να μας πείτε για το πώς μπορούμε να οικοδομήσετε μία γέφυρα με τον ε, διάδοχό σας. Πώς θα... Θυμόμαστε το όνομά του. Όχι, στα σοβαρά τώρα. Φέτος θα είναι η πρώτη φορά που αποφασίσαμε στα πλαίσια των ε, κρατών μελών και του σχετικού κανονισμού να έχουμε το contingent liability σε ό,τι αφορά τους κανονισμούς που υπάρχουν για την ε, δημόσια χρέωση. Υπάρχουν ε, μορφές ε, κρυφής, κρυφού δημοσίου χρέους. Υπάρχει αυτή η σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα που το κινδύνο αναλαμβάνει το κράτος, αλλά στη συνέχεια υπάρχουν προβλήματα, άρα δεν είναι κάποιες επενδύσεις αποδοτικές και ευεργετικές. Γι' αυτό λοιπόν είναι σωστό ότι θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια. Θα θέλαμε λοιπόν να ξέρουμε μέχρι που έχετε φτάσει και πού έχουν φτάσει και τα κράτη-μέλη σε ό,τι αφορά αυτές τις υποχρεώσεις. Εγώ τη βλέπω από τη δική μου χώρα ότι συχνά οι μεμονωμένοι φορείς δεν ξέρουν τι κίνδυνο να λαμβάνουν. Πόσο μάλλον το πώ ε, μπορούν αυτό να το παρουσιάσουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο πληρισμός των χρεών και των ελλημάτων Νομίζω ότι δεν πρέπει να επιτρέπεται να διονύζεται από κρυφά χρέη. Ποια προβλήματα λοιπόν θεωρείτε ότι υπάρχουν ακόμα. Ευχαριστώ. Και ο κύριος Μπάλτς ε, ζήτησε το λόγο, αν δεν κάνω λάθος. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Βίζερ, να επανέλθω σε ένα από τα σημεία που φτάσατε. Στην έκθεση του Ιανουαρίου, την ετήσια έκθεση μάλλον, αναφέρεται ότι ο αριθμός των υψηλής ποιότητας ιδρυμάτων δεν ε, ε, εγγυάται πλήρως το ESS. Πιστεύετε ότι υπάρχει τάση οι στατιστικές υπηρεσίες να μην είναι αρκετά ανεξάρτητες και πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι οι στατιστικές υπηρεσίες θα παραμείνουν ε, υπηρεσίες στατιστικής αξίας και δεν θα πάρουν πολιτική διάσταση. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. Ευχαριστώ. Και τώρα θα ξαναδώσω το λόγο στον κύριο Βίζερ. Για 10 λεπτά παρακαλώ. Για ενδεχόμενα σχόλια και απαντήσεις. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι είμαι πρόεδρος του ΕΣΚΑΠ, του Ευρωπαϊκού Συμφουλίου Φορέα, δηλαδή για τη διακυβέρνηση στον τομέα της στατιστικής. Το G από το ΕΣΚΑΠ, διακυβέρνηση. Εμάς μας απασχολούν περισσότερο μεταζητήματα. Τα μεταδεδομένα, όχι τόσο οι συγκεκριμένοι αριθμοί, τα γυμνά νούμερα. Και παρόλο που σχεδόν όλοι οι συνάδελφοι ε, σχετίζονται με τα στατιστικά θέματα και ήταν προϊστάμενοι υψηλόβαθμοι σε στατιστικές ε, υπηρεσίες ή εθνικά στατιστικά γραφεία, ασχολούμαστε περισσότερο με θέματα διακυβέρνησης. Τώρα, ως προς ερωτήσεις σας. Και κάποιες παρατηρήσεις που κάνατε με έμεσες ερωτήσεις. Μιλήσατε για διορθώσεις διορισμών ή στοιχείων των εθνικών στατιστικών γραφείων. Έχουμε διαδικασία επιλογής και διορισμού των επικεφαλής των Εθνικών Στατιστικών Γραφείων και των ε, υψηλόβαθμων στελεχών που θα πρέπει να είναι αξιοκρατικοί. Και μόνος γνώμονας να είναι τα προσόντα των υποψηφίων σε θέματα στατιστικής. Και όπως και σε άλλες διαδικασίες και εδώ φυσικά υπάρχει α, πλήρης απουσία της εικόνας ότι έχουμε βγάλει τα πιστόλια έξω και περιμένουμε με το πιστόλι στο χέρι. Μερικές φορές είχαμε παρέτηση προϊσταμένων που φαίνεται ότι συμπίπτει όλο τυχαίω με την ανάληψη καθηκόντων νέας κυβέρνησης. Τέτοιες συμπτώσεις τις ε, παρακολουθούμε και σε κάθε περίπτωση εξηγούμε ότι δεν είμαστε ιατροδικαστική μονάδα, ούτε θέλουμε να γίνουμε τέτοια ιατροδικαστική μονάδα, δεν είμαστε ιατροδικαστές και δεχόμαστε καλόπιστα τις εξηγήσεις που μας υποβάλλουν και φυσικά πάντα δίνουμε συστάσεις. Και προσπαθούμε να προλάβουμε την δημοσιότητα. Γιατί θέλουμε πραγματικά αξιοκρατικές διαδικασίες ε, επιλογής και διορισμού στο μέτρο του δυνατού. Τώρα, το θέμα του επηρεασμού των δεδομένων στο θέμα αυτό ή για το θέμα αυτό μάλλον δεν έχουμε καμία απόδειξη και τώρα για τις υπόνοιες ε, το θέμα των ελληνικών στατιστικών έχει διευκρινιστεί οπότε δεν υπάρχουν πια ούτε υπόνοιες για τα θέματα αυτά διευκρίνησε το θέμα της αξιοκρατικότητας που θα πρέπει να χαρακτηρίζει τις διαδικασίες επιλογής δεν έχουμε καμία αμφιβολία για τις δεξιότητες, τα προσόντα, την ακαιρεότητα των διορισμών που γίνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη Eurostat. Στην περίπτωση του κυρίου Ράντεμάχαρ έχουμε ένα ηθήνων στέλεχος και μάλιστα στο φορέα μας, στον ΕΣΓΑΠ, εντυπωσιαστήκαμε όχι μόνο από τις ε, ικανότητες του ως μάνατζερ βασικού διαχειριστεί, αλλά από τις βαθύτατες γνώσεις του για τα στατιστικά θέματα. Θέλουμε και στο μέλλον τέτοιες, τέτοιοι διορισμοί να γίνονται με αξιοκρατικά κριτήρια, επαναλαμβάνω, με βάση τα προσόντα του υποψηφίου, τις δεξιότητες και τις ικανότητές του. Φυσικά κάποιος συνάδελφος την Επιτροπή θα πει αυτό το σύστημα έχουμε, με αυτό πορευόμαστε. Ναι, αλλά θα έλεγα το σύστημα περιτροπής που έχετε δεν εξασφαλίζει ότι ο επόμενος επικεφαλής ε, της Eurostat, γιατί αναπόφευκτα κάποια στιγμή θα αναλάβει κάποιος άλλος. Δεν εξασφαλίζεται λοιπόν ότι ο επόμενος διευθυντής της Eurostat θα είναι εξίσου ε, με τον κύριο Ράντεμάχερ. Βέβαια η Eurostat ε, έχει και ε, με αρμόδια, επιτροπή, ε, στην, με αρμόδια υπηρεσία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Eurostat βρίσκεται στο επίκεντρο του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος. Οπότε θα πρέπει να δώσει το καλό παράδειγμα, να γίνει υπόδειγμα προς μίμηση σε πολλά θέματα. Τώρα, πώς φτάνουμε εκεί, δεν θα ήθελα να περάσουμε σε μια πολιτικοποίηση της συζήτησης. Αυτό αυτός είναι ο κίνδυνος, να είναι πολιτικός ο διορισμός. Ο ρόλος των πολιτικών είναι να εξασφαλίσουν ανεξάρτητη διαδικασία επιλογής και διορισμού. Αυτή είναι η απάντησή μου για το Γενικό Διευθυντή, για την αναλλαγή, για τη διαδοχή του. Και αυτά είχα να πω για τις διαδικασίες πρόσληψης και στελέχωση που θα πρέπει να εξασφαλίζουν ποιοτικού υποψηφίου και σε επίπεδο Eurostat και σε επίπεδο Εθνικών Στατιστικών Ινστιτούτων ή Υπηρεσιών. Ο κύριος Τόρβαλτς ρώτησε πόσο σοβαρά είναι τα προβλήματα. Θα έλεγα ότι κάποια εθνικά στατιστικά Ινστιτούτα έχουμε την αίσθηση ότι παρόλο που δεν εφαρμόζουν κατά γράμμα και ευλαβικά κάθε παράγραφο του κώδικα ορθής πρακτικής, παρόλα αυτά ε, διασφαλίζουν επίπεδο ανεξαρτησίας και δεν δέχονται παρεμβάσεις. Σε άλλες περιπτώσεις έχουμε την αίσθηση ότι οι διορισμοί, οι επαναδιορισμοί, και απογοήτευση, η απόλυση μάλλον, ε, οι απολύσεις κάποιων προϊσταμένων ε, όλος παραδόξως συμπίπτουν με εναλλαγή του πολιτικού κύκλου και της πολιτικής ηγεσία. Πάντως αυτό που θα πρέπει να έχουμε κατά είναι το εθνικό στατιστικό σύστημα δεν αφορά μόνο μία Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, γιατί έχουμε και πολλές περιφερειακές στατιστικές υπηρεσίες. Και όσο κατεβαίνουμε προς την περιφερειακή κλίμακα, προς την τοπική κλίμακα, έχουμε την αίσθηση ότι οι διορισμοί γίνονται με βάση τη εξόδου από την ε, περιφερειακή γραφειοκρατία περισσότερο, παρά με βάση την αξιοκρατία και την καταλληλότητα του υποψηφίου και τα προσόντα του σε θέματα στατιστικής. Αλλά επαναλαμβάνω δεν μιλούμε μόνο για εθνικές στατιστικές υπηρεσίες. Αλλά πάντως δεν θεωρώ ότι το ευρωπαϊκό στατιστικό σύστημα διατρέχει κίνδυνο. Απλώς ε, μερικά εθνικές στατιστικές υπηρεσίες ή μερικά εθνικά συστήματα λειτουργούν καλύτερα από άλλα. Το ίδιο ισχύει και για τη χρηματοδότηση των στατιστικών συστημάτων. Πιστεύουμε ότι η Eurostat ήταν, είναι και θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσει κάποιες δημοσιονομικές περικοπές και μειώσει προσωπικού. Είχαμε πάντως συζητήσει με συναδέλφους ε, επί σειρά ετών και έχουμε και συνομιλίες με τους προϊσταμένους επιλεγμένων εθνικών στατιστικών υπηρεσιών και τους ρωτάμε τι κάνετε με τους σπόρους. Σε κάποιες χώρες υπάρχουν πιέσεις ε, με δυσκολία σε θέματα τέτοια. Αλλά γενικώ θα έλεγα ότι τα δημοσιονομικά προβλήματα δεν ήταν τόσο δυνά στα περισσότερα κρατημέλη για να επηρεάσουν ε, τις στατιστικές υπηρεσίες. Σε μερικές χώρες που έχουν ε, ΑΕΠ κάτω από το κοινοτικό μεσόρο, ίσως σε μερικές από αυτές, δεν θα τις έλεγα πια νέες χώρες μέλη, γιατί έχουν ε, χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί η χρηματοδότηση και το επίπεδο μισθών είναι τέτοιες που δεν εξασφαλίζουν δυνατότητες τελέχωσης πάντα υψηλής ποιότητας. Και έχουμε και διάφορες ερωτήσεις για άλλα ζητήματα, στα οποία δεν θα ήθελα να επισέλθω. Στον κύριο Μπαγιέ θα ήθελα να απαντήσω ότι Οι περισσότερες ερωτήσεις αφορούσαν τη Eurostat και όχι το δικό μας Ευρωπαϊκό Συμβουλευτικό Φορέα. Είναι μόνιμο χαρακτηριστικό της οικονομίας ότι οι επενδύσεις από μόνες τους δεν είναι κατά ανάγκη καλές ή κακές. Οι δαπάνες στην παιδεία, η πρόσληψη δασκάλων είναι φυσικά επένδυση σε ανθρώπινο κεφάλαιο. Βέβαια υπάρχουν αποκλίνωσες απόψεις για το πόσο κοινωνικά παραγωγική είναι μια επένδυση. Αν ενισχύεται με σκυρόδεμα έναν αυτοκινητόδρομο. Πάντως υπάρχουν ορατές και σημαντικές εξαιρέσεις. Για παράδειγμα στο Σύμφωνο Σταθερότητας ε, τις γνωρίζουμε ως οικονομολόγοι ότι ο κόσμος μας είναι ατελής και το, στατιστικό μας σύστημα είναι ατελές. Γι' αυτό και μερικές φορές ε, γίνεται εθνικός χαρακτηρισμός των επενδύσεων. Και αυτό δεν εμφανίστηκε μόνο στο φαινόμενο το 2010, ήταν από το 1995 και θα συνεχιστεί και στο μέλλον. Πιο σημαντικό είναι να επικεντρωθούμε στις οικονομικές προτεραιότητες των κρατών μέλων και όχι στις στατιστικές πληροφορίες αυτές καθ' αυτές. Κύριε Γκίγκολτ, ρωτήσατε για τις υποχρεώσεις και τι γίνεται με τις απρόβλεπτες ανάγκες. Όντως υπάρχουν κάποια κενά εκεί και από το 2010 το σύστημα του 2010 έχει σε κάποιο φως, σε κάποια στοιχεία του παθητικού, σε κάποιες υποχρεώσεις που αφορούσαν κυρίως μη κυβερνητικέ οργανώσεις και οντότητες. Βλέπετε τι άλμα είχαμε στο λόγο χρέος προς ΑΕΠ. Εκεί το χρέος κάποιων οντοτήτων και οργανώσεων ε, υπολογίστηκε στον ιδιωτικό τομέα, ενώ κανονικά ήταν χρέος του δημόσιου. Για παράδειγμα, το χρέος ε, σιδηροδρομικών ε, εταιριών ή νοσοκομείων. Μπορεί να θεωρείται αυτός πρόοδος, αλλά δεν συνιστά κάτι τέτοιο μια στατιστική τελειοποίηση. Τώρα για τις κοινοπραξίες δημοσίου ιδιωτικού φορέα δεν αφορά κάτι τέτοιο τη στατιστική διακυβέρνηση, αλλά περισσότερο τη στατιστική διαφάνεια. Και ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να πω ότι όλα αυτά τα θέματα από κοινού φροντίζουν ε, να, παίζουμε σημαντικό ρόλο ε, ως δείκτες ε, οικονομικής πολιτικής και όχι ως μεταβλητές της οικονομικής πολιτικής. δεν έχουμε μία κοινή κινητήρια δύναμη για τα στατιστικά. Γι' αυτό και θα πρέπει όλο και περισσότερο να χρησιμοποιούμε περίπλοκους κανόνες και υπάρχει κίνδυνος και η ανάγκη να μην χάσουμε το βαθμό εγρήγορσης και απαγρύπνησής μας. Και προσβλέπω και στη δική σας βοήθεια για να ασκούμε αυτή την επαγρύπνηση και την εγρήγορση. Σας ευχαριστούμε κύριε Βίζερ, θα παραμείνουμε σε επιφυλακή και σας ευχαριστούμε για την καλή συνεργασία όλα αυτά τα χρόνια. Ελπίζουμε ότι και με το διάδοχό σας θα έχουμε ε, πολύ καλή συνεργασία. Θα περιμένουμε επίσημες πληροφορίες για να ε, ασκήσουμε και μέσα στις αρμοδιότητές μας και ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία για τον διορισμό τριών μελών από την πλευρά του Κοινοβουλίου. Περιμένουμε τα γραπτά σχόλια των συντονιστών και τα ονόματα θα ανακοινωθούν στους ενδιαφερομένους στη διάσκεψη των Προέδρων. Θα ολοκληρωθεί λοιπόν σύντομα η εξέταση του σημαντικότητα αυτού κανονισμού για τις στατιστικές για να αποσαφινιστούν τα θέματα ε, τα οποία σχολιάσατε και με τα οποία συμφωνώ μαζί σας. Σε δύο λεπτά ψηφίζουμε. Okay, colleagues, Συνάδελφοι, ας ξεκινήσουμε με τις ψηφοφορίες. Να κοιτάξουμε λίγο αν λειτουργεί η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία για έλεγχο. Άρχεται η ψηφοφορία. Ναι, ναι, τεστ κάνουμε, δοκιμή. Ψηφίστε παρακαλώ.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 Κυρία Φερέιρα, πρόεδρε, πριν περάσουμε στις ψηφοφορίες αυτές καθεαυτές, να καταστήσω σαφέστατο το εξή, γιατί δεν δηλώνεται στον κατάλογο ψηφοφοριών ότι για την ομάδα των σοσιαλιστών και δημοκρατών είναι κόκκινη γραμμή. Είναι απαγορευτικό εάν σε συμβαστική α και στη συμβαστική σ, όχι όχι, στη συμβαστική α μισό λεπτό και σ, ναι, Εάν οι όροι αρκεί όλα τα ένομα μέσα προσφυγής κατά της απόφασης αυτής να εξαντληθούν. Εάν αυτό υπερψηφιστεί, ε, είναι για μας κόκκινη γραμμή. Σημαίνει ότι όλες οι διαδικασίες που μπορεί να ε, χρησιμοποιηθούν κατά μιας κύρωσης και εφόσον έχουν εξαντληθεί πριν την επιβολή της κύρωσης, αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει καμία νομική βεβαιότητα. Οπότε δεν έχει κανένα νόημα να προβλέψουν ένα τέτοιο πλαίσιο. Ήθελα να καταστεί απολύτω σαφέ. Με συγχωρείτε που το λέω και το δηλώνω προηγουμένω, αλλά είναι θέμα διαφάνεια και σεβασμού των υπολείπων ομάδων. Για να διευκρινίσουμε αυτό που υπόθηκε. Οι σοσιαλιστέ θεωρούν καθοριστική ψηφοφορία το δεύτερο τμήμα τη συμβαστική A, με μείον δηλαδή. Με πρόσημο μείον. η ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών θεωρούν ε, καθοριστική ψηφοφορία και το, την απόρριψη του, την καταψήφιση του τμήματος 2. Τώρα θα ψηφίσουμε λοιπόν τι εξουσίε τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για επιβολή κυρώσεων. Ξεκινούμε με την τροπολογία 2. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται. 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 4. Υπέρ. Κατά. Καταπίπτει αν εγκριθεί. Αλλά δεν εγκρίθηκε 14, οπότε να ψηφίσουμε και την 4. <coughs> Σωστά, ωραία. Λοιπόν, ψηφίζουμε. Ξανά. 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται νομίζω. Συμβαστική Α με ξεχωριστή ψηφοφορία. Κατά τμήματα μάλλον ψηφοφορία. Πρώτο τμήμα, χωρίς τους όρους που διάβασε και η Ελίζα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τμήμα 2, υπέρ, κατά, νομίζω να ψηφίσουμε ηλεκτρονικός. Άρχεται η ψηφοφορία. Λείπει ένας συνάδελφος. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 19 με προφορική τροποποίηση. Πρέπει να διαβάσω. Διαβάζω την προφορική τροπολογία. την ε, διαδικασία επιβολής κυρώσεων. Αντίρρηση, αντίρρηση στην προφορική τροπολογία. Τέσσερα μέλη έχουν αντίρρηση. Πούντα. Ένας. Χρειαζόμαστε τέσσερις. Δύο. Τρεις. Δεν έχουμε τέσσερις ξαναδιαβάζω την προφορική τοπολογία. Κατά την άσκηση των εποπτικών τη καθηκόντων και τη συλλογή στατιστικών πληροφοριών, η διαδικασία επιβολή κυρώσεων για το Ταμείο Εξυγένσης. Ε, υπέρ, κατά, ελέγχουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Με μία ψήφο διαφορά. Τώρα, αρχική τροπολογία. Επέρ. Κατά. Και πάλι έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Τροπολογία 19 χωρίς την προφορική τροπολογία. Απορρίφθηκε. 20. Κατά τμήματα ψηφοφορία. Τμήμα 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τμήμα 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Τμήμα 2. απορρίφθηκε. Απορρίφθηκε. Πέντε υπέρ. Κατά. Έλεγχος. Πέντε Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 21 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 22 υπέρ. Κατά. Θα ψηφιζόταν μόνο αν είχε εγκριθεί η 21η. Συμβαστική B. Υπέρ. Η 22 μπορεί να ψηφιστεί μόνο αν εγκριθεί η 21η, όχι το αντίστροφο. B. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 8. Υπέρ κατά αποχές νομίζω εγκρίθηκε 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική C κατά τμήματα ψηφοφορία πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές Εγκρίνεται. Πήμα 2. Υπέρ. Κατά. Έλεγχος. Ελέγχουμε και το δεύτερο τμήμα. Και ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 11. Εάν εγκριθεί θα γίνει εξή ε, γλωσσική διορθώση. Έχετε το κοινό, δεν το διαβάζω. Υπέρ, κατά, αποχέ, εγκρίνεται. 12. Υπέρ. Κατά. Έλεγχο. Για την 12. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Εγκρίνεται. 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα ψηφίζουμε το κείμενο στο σύνολό του. Με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Και τώρα ψηφίζουμε το νομοθετικό ψήφισμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Ένα συνάδελφος δεν ψήφισε. Πέρας. Έτσι κι αλλιώς. Εγκρίνεται. Μηδέν. Αποχές 31 ψήφι υπέρ, 24 Και τώρα περνάμε Στη δεύτερη έκθεση. Συλλογή στατιστικών πληροφοριών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Τροπολογία 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Αγκρίνεται. 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Αγκρίνεται. 6. Με προφορική τροπολογία. May αντί για δύνατε αντί για πρέπει. Υπέρ, κατά, αποθές, αγκρίνατε. Επτά, αποσύρετε, οκτώ, υπέρ, κατά, αποθές, αγκρίνατε. Εννέα, υπέρ, κατά, αποθές, αγκρίνατε. Δέκα, υπέρ, κατά, Έλεγχος για την τροπολογία 10. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται η τροπολογία. Μια 11 και 12 αποσύρονται. 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. 14. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 15. Αποσύρεται. 16. Υπέρ κατά έλεγχος για την 16 άρχεται την ψηφοφορία. Πέρας, απορρίπτεται. 17 υπέρ, κατά. Νομίζω η ίδια πλειοψηφία έχει δημορφωθεί. Για να το ελέγξουμε το 17. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 18 με τεχνική διόρθωση. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 19 και 20 αποσύρονται. Πρώτη. 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ηλεκτρονική ψηφοφορία για το κείμενο όπως τοποποιήθηκε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 48 υπέρ, 6 κατά, 2 αποχές. Τώρα ψηφίζουμε το νομοθετικό ψήφισμα. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρασε. 48 υπέρ, 8 κατά. Η έκθεση, η έκθεση εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στους δύο εισηγητές. Και ε, η συνεδρίαση λίγη. Στις 3 θα ξαναρχίσουμε.